Bonjour à tous. Buenos días. Καλημέρα σα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνεδρίαση. Υποχρεωτικά πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρα πολύ αποσχολημένο πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε και μια κοινή συνεδρίαση, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στις 10 και 4 νομίζω ότι ε, έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν να έχετε μαζί σας και τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Αν όχι, στείλτε κάποιον να σας τη φέρει. Και θα έρθει και η Επίτροπος Vivian Ρέντινγκ για να μα πει για το πρόγραμμα εργασία από το 2013 και τούδε στον τομέα τη δικαιοσύνη. Θα έρθει στι 11 περίπου και θα μείνει μέχρι τι 12 και 4 και κατόπιν έχουμε συνεδρίαση συντονιστών. Ένα σύντομο διάλειμμα στι 2. Έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση στη συνέχεια. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών οργανώνει μια ακρόαση για την κατάσταση στην Ουγγαρία κατόπιν αιτήματο κάποιων πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των φιλελευθέρων και των πρασίνων και η ακρόαση θα διαρκέσει δύο ώρες και ένα τέταρτο. Μας περιμένει λοιπόν πολλή δουλειά σήμερα και σας το λέω γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το χρονοδιάγραμμα. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο παριθμών 1 για το σημείο 6 τώρα της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Κοέλιο, ο εισηγητής, πρότεινε να αναβληθεί η ψηφοφορία επιβεβαίωσης που είναι προγραμματισμένη για σήμερα για την έκθεσή του, επομένως δεν θα γίνει. Εάν δεν υπάρχει καμία ένσταση λοιπόν, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και επίσης να σας ανακοινώσω ότι οι συντονιστές ενέκριναν τους ακόλουθους εισηγητές ε, για το δικαιοσύνη 10 τον κύριο Φιλ Κλέης. Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας Συνόρες, ο κύριος Μόλτερ. Προστασία των πολιτών ε, σε προξενικό επίπεδο ε, για πολίτες στο εξωτερικό, Edith Bauer. Πρόγραμμα προστασίας στο ευρώ κατά της ε, παραποίησης, ο κύριος Αγουστίν Διασδεμέρα. Πρόγραμμα Ιθαγένειας, κυρία Κίνγκα Γκάντς. Και αλλάγησε και ο εισηγητής στον ε, κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Γενικές Διατάξεις για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και το σχετικό ταμείο. Η έκθεση είχε δοθεί στον κύριο Λορένσο Φοντάνα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κύριο Μάριο Μποργκέτσιο για την ομάδα των συντηρητικών και δημοκρατών. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις λοιπόν εγκρίνονται και αυτά και περνάμε στο πρώτο σημείο κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Γυναικών. Και για άλλη μια φορά λοιπόν, έχω τη χαρά να καλωσορίζω εδώ τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Είναι και ο πρόεδρος, ο κύριος Γκούσταυσον. Καλωσορίσατε. Είναι τιμή μου να συμπροεδρεύω μαζί σας ε, για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Το σχέδιο έκθεσης δηλαδή για την οδηγία που καθορίζει ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Έχουμε δύο εισηγήτριες, η Τερέσα Χιμένε Πεθερίλ Λμπάριο και η κυρία Αντώνια Παρβανόβα. Και να σας υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που θέλει να ενισχύσει τα δικαιώματα των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε το Μάιο του 2011 και έχει ακολουθηθεί η συνήθιση νομοθετική διαδικασία. Είναι συναρμόδιες οι επιτροπές, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Γυναικών και ε, συνεργάζονται βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού. Here. Thank you. Article 51 Uh, το Δεκέμβριο το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγιση ώστε η Δανική Προεδρία να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Uh, draft report. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό σχέδιο έκθεση των δύο επιτροπών, το οποίο αντανακλά τη συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητριών και θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών εκπνέει στις 27 Φεβρουαρίου. By noon, 1200. Στις 12 το μεσημέρι. Οι τροπολογίες θα εξεταστούν στις 21 Μαρτίου, ψηφοφορία στις 27 Μαρτίου και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκούσταυσον, πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, για να σχολιάσει και να κάνει παρατηρήσεις και κατόπιν θα ακούσουμε τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Χιμένες Μπεθερίλ και την κυρία Παρβανόβα, οι οποίες θα μας παρουσιάσουν τα στοιχεία της έκθεσης. Will have an to take the floor, Και από εκεί και πέρα θα δώσουμε το λόγο και στα μέλη. Κύριε Γκούσταυσον. Ευχαριστώ και είναι μεγάλη μου τιμή που συμπροεδρεύω με τον κύριο Αγγιλάρ. Θα μιλήσω σου ειδικά εγώ. Σας παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας για να με καταλάβετε. Είναι πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία των δύο επιτροπών. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας αυτό. Ε, και για αυτές τις εκθέσεις και μιλώντας εξ ονόματος της Επιτροπής των Γυναικών ε, πρόκειται για εκθέσεις ε, ιδιαίτερης βαρύτητας διότι κάνουμε παρεμβάσει έχοντα κατά νου το θέμα της ε, ισότητας των δικαιωμάτων των δύο φύλων και ξέρετε ότι επηρεάζεται η κατάσταση των γυναικών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τις γενικέ κατευθυντήριες γραμμές της κυρίας Χιμένη και της ε, κυρίας Παρβάνοβα. Ε, επίσης, ε, υποστηρίζουμε σε κάποιο βαθμό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σίγουρα επιδέχεται πάρα πολλές βελτιώσεις σε αυτή η αρχική πρόταση. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για ένα γενικό ορισμό της έννοιας του θύματος. Προσπαθούμε να ε, θεσπίσουμε ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την διερμηνία, την ενημέρωση, την νομική αρρωγή και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν γίνει πολύ καλές προτάσεις από τις δύο εισηγήτριες, ε, διότι δίνουν μια βασική δυναμική στο θέμα της προστασίας των θυμάτων και αναφέρονται σε δύο βασικά ε, ζητήματα, παραδείγματο χάρη η βία που σχετίζεται με το φύλλο και θυματοποίηση των γυναικών. Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι με αυτή την επικοδομητική συνεργασία τελικά θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτές τις δύο τόσο σημαντικές εκθέσει. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκούσταυσον. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τις συζητήτριέ μας. Η κυρία Χιμένη Βασαρίλ θα αρχίσει και στη συνέχεια η κυρία Παρβάνοβα. Θα ήθελα αν συμφωνείτε να μιλήσετε για πέντε λεπτά, όχι παραπάνω, για να προλάβουμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών. Έχουμε πάρα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα και το λογικό ίσως θα ήταν δύο λεπτά έκαστη, γιατί έχουμε και την ψηφοφορία και ξέρετε ότι στις ψηφοφορίες έχουμε συμπρογραμματίσει με άλλες επιτροπές, έρχονται ε, συνάδελφοι, δεν έχουν χρόνο. Τέλος πάντων πρέπει να είμαστε ακριβείς με το χρονοδιάγραμμα στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Είναι για μένα τιμή να είμαι συγγήτρια, συνεισηγήτρια εξ ονόματος Επιτροπής μας με την κυρία Παρβάνοβα. Είμαι μέλος και στις δύο επιτροπές και είχα την ευκαιρία να, να παρακολουθήσω συγγνώμη, πολλές εκθέσεις σε σχέση με τα θύματα και λόγω της προσωπικής μου ζωής έχω ζήσει στην ε, ζωή μου και στην οικογένειά μου. Η τρομοκρατική οργάνωση η ΕΤΑ ε, στη Σεβίλη δολοφόνησε τον αδελφό μου και την ύφη μου. Είναι λοιπόν κάτι που με αφορά προσωπικά. Όταν άρχισα να ασχολούμαι αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσα ότι η μεγάλη ξεχασμένοι σε αυτή την υπόθεση είναι τα θύματα. Το αντίθετο θα πρέπει να συμβαίνει. Και πραγματικά είναι μία από τις εκθέσεις που τιμούν ε, την εργασία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέθεσε αυτή την πρόταση και την ε, εισηγήτρια κυρία Παρβάνοβα τη Γραμματεία και όλες τις οργανώσεις στήριξης των θυμάτων που συνεργάστηκαν μαζί μας. Ακριβώς επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα και είμαι πολύ δεσμευμένη στην κατεύθυνση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση να επιβληθούν ελάχιστα πρότυπα σε όλη την Ένωση. Και είμαι πεπισμένη ότι η Δανική Προεδρία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ προ την κατεύθυνση αυτή για να βρούμε και να αναζητήσουμε καλύτερε ε, λύσει ε, σε αυτέ ε, τι εποχέ τη κρίση που είναι αμήλικτε οι περικοπέ. Θα πρέπει να μειωθεί το κόστος και μειώνεται με την ε, αποφυγή της διπλής θυματοποίησης και της προστασίας των θυμάτων. Έτσι εξοικονομούμε υπηρεσίες που εκ των υστέρων θα πρέπει να παρέχονται και είναι πολύ πιο δαπανηρές τα θύματα υποφέρουν, πλήττονται γιατί δεν έχουν εγγυημένα δικαιώματα. Χρειάζεται ενό σύστημα δικαιοσύνης με διαφάνεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα επιγόντω για να ε, πληρωθεί το πρόγραμμα της ε, Στοχόλμη και να δημιουργηθεί ένας χώρος ελευθερία, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν προστατεύονται μόνο τα θύματα και οι οικογένειές τους με στήριξη και προστασία, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα εθνικά δικαστικά του συστήματα, αλλά και σε εκείνα των γειτόνων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ως σημαντικότερο δικαίωμα το δικαίωμα στην πληροφόρηση, άρθρο 4, το δικαίωμα στη διερμηνία και τη μετάφραση, άρθρο 6, το δικαίωμα πρόσβαση στι υπηρεσίε στήριξη θυμάτων, άρθρο 7, το δικαίωμα να γίνονται ε, ακουστά και να ακούγεται τη φωνή τους σε άλλα άρθρα 11 ε, και στο άρθρο 20 ε, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τις ανακρίσεις και την έρευνα. Όλα τα θύματα, ανεξάρτητα από τη ζημία που υπέστησαν, από που προέρχεται η βία ή το επίπεδο της ζημίας, θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την οδηγία. Η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλές φορές δεν ε, καταγγέλουν μια αξιόπινη πράξη στα θύματα γιατί ε, φοβούνται. Έχουν έλλειψη εμπιστοσύνη, είναι ευάλωτα και έχουν τεράστιες πιέσεις. Επίσης είναι πολύ δύσκολα τα νομικά εμπόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ε, τα θύματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και κυρίως σε γλώσσα που να καταλαβαίνουν. Σε ό,τι αφορά τα πιο ευάλωτα θύματα, κατανοούμε αυτό που λέγεται, αλλά θα θέλαμε να χαρακτηριστούν θύματα με ε, ιδιαίτερες ανάγκες. Γιατί δεν τους αρέσει αυτή η έκφραση ότι είναι ευάλωτοι άνθρωποι. Γίνεται λόγο συγκεκριμένα ε, για ε, παιδιά και άτομα με αναπηρία ως πιο ευάλωτες κατηγορίες. Όταν όμως γίνεται λόγος για θύματα με ιδιαίτερες ανάγκες, δεν πρόκειται μόνο για θύματα σεξουαλικής βίας ή δουλεμπορίου, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, ομάδες θυμάτων, όπως είναι τα θύματα τρομοκρατίας που θέλαμε να συμπεριλάβουμε, οργανωμένο εγκλήματος, ε, ε, θύματα Βία με βάση το φύλλο. Όλα αυτά είναι στις ε, τροπολογίες 69, 70 και 71 και 72. Στα θύματα της τρομοκρατίας θεωρούμε ότι κάθε τρομοκρατική δράση θεωρείται προσβολή και επίθεση στους πυλώνες της δημοκρατίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Γι' αυτό θέλουμε ειδική στήριξη και είναι ζωτική σημασία να υπογραμμίσουμε ότι εκείνοι που παραβιάζουν τα ε, δίκαιο προσβάλλοντας ατομικά δικαιώματα ε, επιτίθενται σε συλλογικά δικαιώματα των πολιτών. Τέσσερα θεμελιώδη δικαιώματα ε, που ζητούν τα θύματα. Δικαίωμα ε, στην αλήθεια, στη μνήμη, στη δικαιοσύνη και στο σεβασμό. Γίνονται δεκτά τα δικαιώματά τους και αναγνωρίζονται πριν, κατά και μετά τη ε, δικαστική διαδικασία και την ποινική δίκη. Είναι πολύ δύσκολο να συνεργάζονται οι διοκτικές αρχές, η αστυνομία, ε, οι δικαστές οι εγγελής θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν τα θύματα σύμφωνα με την αξιόπινη πράξη. Γι' αυτό ε, θέλουμε το άρθρο 24 για τη γενική εκπαίδευση και ενημέρωση και κατάρτιση των υπαλλήλων να εφαρμοστεί. Ε, δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι θα βελτιώσετε με το τι τροπολογίε σα στο κείμενο και θα καταλήξουμε σε μια έκθεση δίκαιη, ρεαλιστική που θα ανταποκρίνεται στι θεμητέ προσδοκίε, όχι μόνο των θυμάτων αλλά των πολιτών, όλων των πολιτών που δυστυχώ από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να περάσουν αυτή τη λεπτή διαχωριστική γραμμή και να γίνουν θύματα. Σα ευχαριστώ και πάλι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξή τη, για το Συμβούλιο που θα το ακούσουμε επίση. Ε, τους ε, βοηθούς, τη γραμματεία, τους υπαλλήλους και βεβαίως τη ε, συνεισηγήτρια που ε, τόσο αρμονικά δουλέψαμε μαζί. Ευχαριστώ και σας για τη μελλοντική σας συμβολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιμένες Μπεθερήλ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Παρμανόβα. Αν μπορέσετε να διατηρήσετε κι εσείς πέντε λεπτά θα ήταν εξαιρετικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Χιμένες για την εξαιρετική συνεργασία και να αναγνωρίσω ότι η μέθοδος εργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών ήταν εξαιρετική. Και αυτό λογικά θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και για το Συμβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο γραμματείες των Επιτροπών. Η υποστήριξή τους και η πυρογνωμοσύνη του ήταν εξαιρετικέ και νομίζω ότι συνεισέφεραν ιδιαίτερα στη ποιότητα τη εκθεσή μα. Χρησιμοποίησαμε επίση ε, και ε, υποστήριξη από εμπειρογνώμονε, έγινε ακρόαση και χρησιμοποίησαμε και τι αναλύσει του και είχαμε υποστήριξη και από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω αυτό στη συνέχεια να μα επιτρέψει να βρούμε έναν εύκολο τρόπο ώστε να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των θυμάτων ε, εγκληματικών πράξεων. Σίγουρα το πλαίσιο αυτό θα βοηθήσει ώστε όλα τα θύματα ε, εγκληματικών πράξεων να μπορούν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω ότι δυστυχώς το πρώτο κείμενο που είχαμε ε, ήταν για τα δικαιώματα των ενόχων. Τα θύματα έρχονται στη δεύτερη θέση, αλλά ελπίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το έργο αυτό και μέσω της εκθεσής μας με την κυρία Χιμένες ε, ε, είχαμε ένα κοινό στόχο, να έχουμε ένα κατάλληλο ορισμό για το θύμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ληφθεί υπόψη ο ορισμός αυτός όταν θα σχεδιάζονται οι κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και θα επιμορφώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα θύματα. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα και τρει προτάσει προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχο αυτό. Πρώτον, να έχουμε ένα κατάλληλο ορισμό για το θύμα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καταλήλω στι ανάγκε του. Πριν εισηχθούν νέε διατάξει, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε του ορισμού και τι έννοιε που αναφέρονται στην οδηγία. Δεν θέλουμε να έχουμε νέε ή ξεχωριστέ κατηγορίε θυμάτων, αλλά θέλουμε να έχουμε ένα ξεχωριστό ορισμό που θα μα επιτρέπει να κάνουμε την κατάλληλη αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων. Ω συνεισηγήτρια, θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διάσταση του φύλου στον ορισμό του θύματο και έχουμε και έναν ορισμό για τη βία ε, βάση φύλου στο άρθρο, στην τροπολογία 31. Ορισμένες φορές έχουμε ε, επιθέσεις κατά ανθρώπων λόγω του φύλου τους και ορισμένες φορές αυτές οι μορφές επίθεσης ε, αφορούν γυναίκες. Το 1 τέταρτο όλων των γυναικών έχουν ε, ζήσει ή έχουν υπάρξει θύμα σωματικής βίας και ε, πάνω από ένα όγδο έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Υπάρχει και η τροπολογία 32 για να Έχουμε ε, τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν από ε, συντρόφους, πρώην συντρόφους ή μέλη της οικογενείας και εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει λυπής προστασία των θυμάτων. Επίσης μας ενδιαφέρει η αναφορά σε θύματα τα οποία ε, ε κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό ε, λόγω εκφοβισμού ή είναι κατά επανάληψη ε, θύματα βίας. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις των ε, ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες που ανέφερε η κυρία Χιμένες και μας ενδιαφέρουν οι τροπολογίες 63, 64 και 67 για το θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι ο όρος ευάλωτος έχει αρνητικές προεκτάσεις και ορισμένες φορές πολλά θύματα δεν θέλουν να θεωρούνται ότι είναι ευάλωτα, αλλά ω άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία. Ε, δεν θα θέλαμε να τους εντάξουμε στην ίδια κατηγορία. Επίσης, έχουμε αναφέρει τα θύματα ε, στη νέα κατηγορία των ιδιαίτερων αναγκών, τα θύματα που έχουν ε, υποστεί επίθεση λόγω του φίλου τους Επίσης υπάρχουν κάποια θύματα τα οποία ε, θεωρούνται ότι έχουν ιδιαίτερε ανάγκες, γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να τους προστατεύσουμε κατά νέλος και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται σε προσωπικό επίπεδο αναπερίπτωση και να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπω η ηλικία, το φύλλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμό, η φύση του εγκλήματο και κατά πόσον είναι αλλοδαπό το θύμα. Επίσης ε, θα πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόζονται καταλήλως τα μέτρα για όλα τα θύματα. Υπάρχουν ε, νέοι ορισμοί στο άρθρο 18α για υπηρεσίες ε, προστασίας των θυμάτων που λαμβάνουν υπόψη τους και τη διάσταση του φύλου, την ισότητα του, των, μεταξύ των φύλων και θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό για να μην υπάρχει και σε δεύτερο επίπεδο θυματοποίηση. Υπάρχει το άρθρο 18β το οποίο προσφέρει συνδρομή σε θύματα σεξουαλικής βίας όπως επίσης παροχή ε, στέγης, ε, ψυχολογική και νομική συνδρομή ε, και λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα των θυμάτων λόγω Υπάρχει και πρόβλεψη για κατάλληλη επιμόρφωση των ανθρώπων που θα έρθουν σε επαφή μαζί τους, όπως για παράδειγμα αστυνομικών, και να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη για θύματα με συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαίτερα θύματα βίας λόγω φύλου ή βίας ε, μέσα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Θεωρούμε επίσης ότι η επιμόρφωση και η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να γίνεται σε στενή διαβούλευση και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με υπηρεσίες για προστασία θυμάτων ε, που έχουν υποστεί ε, βία λόγω του φίλου τους και θα πρέπει αυτό να γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τα συμπληρωματικά μέτρα για την προστασία των θυμάτων, για την κατάλληλη πρόληψη, Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί οποιαδήποτε νέα δομή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρχών, ο οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση των θυμάτων και έχουν εντοπιστεί εξή κατηγορίε. Βοήθεια προ τα θύματα, συλλογή δεδομένων, Υπάρχουν ε, ήδη ευρωπαϊκέ οργανώσει που ασχολούνται με τι ανάγκε των θυμάτων. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο παρατήρηση και βοήθεια προ τα θύματα και θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία που θα λαμβάνει και στοιχεία όπω η ηλικία και η εθνικότητα των θυμάτων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, συλλέγονται περισσότερε πληροφορίε και να υπάρχουν και κατάλληλε εκστρατείε ενημέρωση ώστε τα θύματα να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα επιπλέον μέτρα τα οποία προτείνουμε στην πρότασή μας μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις νέα κατανομή πόρων ή κάποια αύξηση, αλλά όχι και τόσο πολύ αύξηση, αλλά νέα ε, κατανομή των πόρων ώστε να πάνε στις κατάλληλες αρχές. Θα πρέπει να υποθυμίσουμε βεβαίως ότι όπως εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό κόστος των εγκληματικών πράξεων, όχι μόνο για τα θύματα, αλλά και για το κράτος και την κοινωνία στο σύνολό τη, εκτιμάται στα 233 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και αυτό δεν προκύπτει μόνο από τις εγκληματικές πράξεις, αλλά και από το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη προς τα θύματα για να μπορέσουν να ε, αντιμετωπίσουν τις δικαστικές διαδικασίες και να συνέλθουν και επομένως θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά και θα μπορέσουν ε, να βοηθήσουν ώστε να καταγγέλλονται τα εγκλήματα και να βοηθούνται τα θύματα και μέσω των συστημάτων δικαιοσύνης και μέσω των συστημάτων υγείας. Αυτά είναι τα μέτρα λοιπόν που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι με τα μέτρα τα οποία θα προτείνουν και οι συνάδελφοι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την έκθεσή μας και να έχουμε μια ισχυρή θέση για το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Τώρα Κανονικά θα πρέπει να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θέλω να λάβουν το λόγο. Σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε κατάλογο μιλητών που θέλουν να βάλουν το λόγο και έχουμε και χρονικούς περιορισμούς. Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Άλεν, Άλτεν. Άλεν, Άλτεν, πώς λέγεστε, κύριος, κυρία. That's Mr. Άλτεν, Άλτεν. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Δεν πρόκειται να σχολιάσω κάποιε επιμέρου τροπολογίε. Θα ήθελα μόνο να σα ε, διευκρινίσω ποια είναι η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι έχει γίνει στι μέχρι τούδε συζητήσει. Βασίζεται η πρότασή μα ε, στι ανάγκε των θυμάτων και στην κάλυψή του. Ε, αναγνωρίζουμε τις πέντε ανάγκες, αξιοπρεπή μεταχείριση, υποστήριξη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αντι, ε, επανόρθωση και αποζημίωση. Και σίγουρα η έκθεση ακολουθεί την ίδια γραμμή. Είναι πάρα πολύ θετικά τα στοιχεία που εμπεριέχει και πολύ καλές τροπολογίες. Ε, υιοθετήσαμε την εξή προσέγγιση. Ο σκοπό μα ε, είναι να καλύψουμε όλα τα θύματα αξιόπινων πράξεων. Θέλουμε να μεριμνήσουμε ούτω ώστε κάθε μονομένη περίπτωση να τύχει ε, τη κατάλληλη μεταχείριση. Ταυτόχρονα ταξινομούμε σε διάφορε κατηγορίε τα θύματα και να γνωρίζουμε ότι έχουμε διαφορετικέ ανάγκε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ισορροπία την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια τη διαδικασία θα προσδιορίσουμε αυτέ τι ειδικέ ανάγκε και θα επιτύχουμε αυτή την επιθυμητή η ισορροπία είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μην παραμελήσουμε ή να μην είναι, έχουν πιο προνομιακή θέση κάποια θύματα ε, βάσει των διατάξεων της οδηγίας. Έχουμε ισχυρές φιλοδοξίες, βεβαίως ζούμε αυτή την ε, οικονομική κρίση, όπως σωστά είπαν οι κυρίες Χιμένες, Μπεσερίλ και Παρβάνοβα ενδεχομένως θα έχουν δημοσιονομικό κόστος οι προτάσεις αλλά επίσης θα μειώσουν γενικότερα το κόστος ε, των αξιόπινων πράξεων ε, για την κοινωνία ε, γενικότερα. Θέλουμε πάντως, ακόμη και στο τελικό σχέδιο της έκθεσης, να έχουμε ένα μεν φιλόδοξους στόχους, αλλά και εφικτούς, ρεαλιστικούς. Ε, ως προς το αν μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο, κυρίω ω προ την ισότητα των δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, φρούδες ελπίδες. Θέλουμε ε, να ε, είναι ρεαλιστικά αυτά που προτείνουμε, εφικτά επιτόπου, εφαρμόσιμα και επίση θέλουμε τα ίδια τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, α έχουμε κατά νου ότι οτιδήποτε προτείνουμε ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω νομοθετημάτων ε, και ενδεχομένως κάποια μέτρα θα μπορούσαν να ε, εφαρμοστούν μέσω πιο πρακτικών μέτρων, εφαρμοστικών δηλαδή διατάξεων στο μέτρο του δυνατού. Προσπαθούμε οι προτάσει μας να είναι όσο των δυνατόν ακριβέστερε γίνεται από νομοθετική, νομοτεχνικής, συγγνώμη, νομοπαρασκευαστική πλευράς. Και θα πρέπει να προσέξουμε επίση τη διατύπωση για λόγου εφαρμογή, ε, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώ ποιε είναι οι υποχρεώσει του και άρα βασικό μα μέλημα είναι οτιδήποτε προτείνουμε να είναι ακριβέ και εύληπτο στο μέτρο του δυνατού. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ε, να παραμείνουμε στο πεδίο του άρθρου 82, γιατί αυτή είναι η νομική μας βάση. Η τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι συγγήτριες είναι ιδιαίτερα θετικές και συνιστούν πολύ σημαντικό εφαλτήριο για τις μελλοντικέ συζητήσεις. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα εκπρόσωπος του Συμβουλίου, Όλμερ, από πλευρά της Δανικής Προεδρίας. Δύο λεπτά έχετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ακούσαμε την παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης. Πρόκειται για ένα σχέδιο καταλητικής σημασίας για την εφαρμογή του προγράμματος ε, της Στοκχόλμης και συνιστάμε μεγάλη προτεραιότητα ε, για την Προεδρία μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε τι εργασίε του, ώστε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα και την προστασία των θυμάτων. Είμαι δε πεπισμένο ότι επί Δανική Προεδρία θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, ε, το Συμβούλιο είχε εργαστεί εντατικά, επεξεργαζόμενο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν το Δεκέμβριο. Καταλήξαμε σε μια κοινή θέση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Χιμένες Μπεσερίλη και Παρβάνοβα για την έκθεσή τους η οποία ενέχει ουσιαστικότατες ε, προτάσεις ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα τις εξετάσουμε εκ του Σύνεγγης. Επίσης, η έκθεση τονίζει πως η προστασία των θυμάτων είναι ένα θέμα που θεωρείται προτεραιότητα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχοντας ακούσει την ε, σημερινή παρουσίαση αυτή της έκθεσης, διαπιστώνω με μεγάλη μου χαρά ότι σε διάφορους βασικούς τομείς του σχεδίου είναι παρεμφερείς οι ιδέες και οι προσεγγίσεις που υιοθετούμε. Αληθεύει επίσης ότι υπολείπονται κάποια ε, σημεία που εκκρεμούν που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στο μέλλον. Όμως ε, είμαι και εγώ πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο πριν πριν η Προεδρία μας. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ σύντομα στις διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο απηχούν αυτές τις διαπραγματεύσεις τι επιθυμίες των κρατών μελών. Δηλαδή, την επιθυμία συγκεκριμένα να έχουν μια οριζόντια οδηγία που θα κατοχυρώνει επαρκή προστασία για τα θύματα αξιόπινων πράξεων. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό για το Συμβούλιο το εργαλείο αυτό να είναι αποτελεσματικό και να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη κυρίως από πλευράς του Συμβουλίου διατηρήσαμε το σημείο κίνησης, αν θέλετε, το εφαλτήριο της Επιτροπής ε, του Τέστην, όχι τις μεμονωμένες ανάγκες ε, των θυμάτων που εκείνες θα προσδιορίζαν την αρρωγή ε, από πλευράς των κρατών μελών. Στο Συμβούλιο η θέση μα έχει ω εξή. Αναγνωρίζουμε ότι κάποια θύματα, κάποιε κατηγορίε θυμάτων έχουν συγκεκριμένε και πολύ ειδικέ ανάγκε προστασία. Ω εκ τούτου, κρίναμε πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε μέσα στην έκθεση ότι οφείλουμε να κάνουμε μία κατά περίπτωση αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων και άρα η προσέγγιση μας ε, δεν είναι ε, προσδιορισμένη εκ των προτέρων αλλά αναλύεται κατά περίπτωση. Θα συνεχίσουμε την εξέταση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο όλων των δυνατοτήτων ε, ειδικότερη υποστήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε σε κάποια θύματα ε, σε συνάρτηση με τι ειδικέ του ανάγκε. Όπω σα έλεγα, για το Συμβούλιο είναι επίση ε, σημαντικό, απαραίτητο θα έλεγα, να ε, μην υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στα δικαιώματα των θυμάτων και το δικαίωμα ε, δικαιωρικής υπεράσπισης. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η κεντρική ιδέα της έκθεσης ε, του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο. Θεωρεί επίσης, όπως σας έλεγα, ότι θα πρέπει να είναι ευχρήστο, εύληπτο και ευεφάρμοστο το σχέδιο αυτό στην πράξη. Ε, θα πρέπει να είναι σαφέστατα προσδιορισμένα τα δικαιώματα των θυμάτων, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται ταυτόχρονα ευελιξία η οποία θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε στην πράξη ρεαλιστικές λύσεις. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικονομική συγκυρία από αυτή την πλευρά. Είναι ένα σχέδιο οδηγίας ε, που θεσπίζει μήνυμης ε, πρότυπα, άρα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν αυτά τα πρότυπα εάν το επιθυμούν. Κλείνοντας να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που με προσκαλέσατε στι συνεδρία. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις που καταθέσατε και εξ ονόματος Δανικής Προεδρίας ε, με μεγάλη χαρά θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με τις κυρίες ε, Χιμένες Μπεζερίλε και Παρβάνοβα. Ευχαριστώ την Κομισιόν και την Προεδρία. Ανοίγει η συζήτηση. Δύο λεπτά έκαστος, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Η κυρία Γκρισμπέκ έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ένα δίλεπτο τι να πω. Προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να χαιρετήσω και πάλι την πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ καλή αυτή η μέθοδος των μεικτών επιτροπών που ε, τρέπει να ε, έχουμε πιο εύστοχη και πιο συστηματική δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο συγκίτριες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το θέμα αυτό της ελάχιστης προστασίας των ελάχιστων προτύπων για την προστασία των θυμάτων. Συμφωνούμε λοιπόν σχεδόν με όλες τις ε, προτάσεις των εισηγητών, των εισηγητριών καλύτερα που μόλις μας παρουσίασαν. Θα κάνουμε όμως και μερικές τροπολογίες ε, για μερικές προσθήκες που έχουμε για το κείμενο. Βεβαίως είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια ισορροπία δηλαδή από τη μια να έχουμε τη δίωξη των ε, υπευθύνων και την προστασία από την άλλη των θυμάτων. Στην έκθεση αυτή χαίρομαι ε, για την προσπάθεια που γίνεται για την προστασία των θυμάτων. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο το υπόδειγμα, το πρότυπο κράτους δικαίου ε, που ε, κυριαρχεί στην Ένωση. Θα πρέπει λίγο να στρέψουμε το φως και την προσοχή μας στα δικαιώματα των ε, θυμάτων δεν εστιάζουμε συχνά στα θύματα. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες, ε, στην ευάλωτη φύση των θυμάτων. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι μόνο να διώκουμε τους υπετίους, αλλά να ε, προστατεύουμε τα θύματα, να τα ενημερώνουμε, να τα υποστηρίζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο. Ακόμα και αν είναι δύσκολο αυτό, ακόμα και αν η οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ε, μπορούν τα θύματα να βρίσκουν το δίκιο τους Έχουμε λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση θελησιοκρατική, ε, βολονταριστική, βοήθεια των ε, θυμάτων και εις μεταχείρισης, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω μερικά στοιχεία ε, επιπλέον προστασίας που θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε. Για τις ευάλωτες κατηγορίες προσώπων, κυρίως τα παιδιά, ε, οι ανακρίσει ή ακροάσει μάλλον των ανηλίκων θυμάτων θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο από ε, ειδικού επαγγελματίε που έχουν καταρτιστεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ε, αυτό είναι και το άρθρο 24 που κάνει λόγο για την επιμόρφωση των υπαλλήλων να γνωρίζουν ιδιαίτερα τα θέματα της βίας με βάση το φύλλο και να έχουν αντίστοιχες και αρμόσες συμπεριφορές. Επίσης, καινοτομία, ανταλλαγή εμπειριών είναι χρήσιμες και ε, δίκτυα και υποδομές. Έχω και άλλα πολλά να πω, αλλά τι να κάνω στις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Ε, Τρία. Πρώτον, εγώ είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι είναι ζωτική σημασία στο γεγονό ότι αναφέρονται και τα δικαιώματα των, ε, των γυναικών, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι αυτό είναι το μόνο σημείο στο οποίο ασχολούμαστε με τα ε, θύματα γυναίκε, ε, θύματα σεξουαλική βία, ε, ακροτηριασμού γενετικών οργάνων κ.ο.κ. Ε, υπάρχουν και άλλε περιπτώσει στι οποίε θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά συνολικά. Δεν θα πρέπει να το λησμονούμε λοιπόν αυτό. Δεύτερον, μας χαροποιεί ιδιαίτερα ε, το θέμα των τροπολογιών 53 και 54 για την πρόσβαση σε υποστήριξη και τη δυνατότητα να ε, κάνει κάποιος ε, καταγγελία στην αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα για τα θύματα ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Δεν θα πρέπει δηλαδή να απαγορεύουμε σε κάποιον ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, για παράδειγμα, γιατί δεν έχει τα κατάλληλα έγγραφα για παραμονή σε μια χώρα, να μην έχει πρόσβαση σε προστασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την τροπολογία 54. Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν κάποιοι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συνδικάτα και ούτω καθεξής, για να υποστηρίξουν κάποια θύματα. Δεν θα θέλαμε η οδηγία αυτά να αντιβαίνει ε, με άλλα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε οδηγίες όπως έχουν ε, ε, εγκριθεί στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τα θέματα για την ισότητα και τη σχετική οδηγία. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε. Η οδηγία αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα ως θύματα και αναφερόμαστε και σε θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει Βάλλον. Υπάρχουν και άλλες οδηγίες όπου έχει ληφθεί υπόψη αυτό και το γεγονός ότι αναφέρεται και το περιβάλλον αποτελεί εγγύηση για τη δίωξη θυμάτων, ε, για την συγγνώμη, προστασία θυμάτων όταν υπάρχει θέμα ε, περιβάλλοντος. Θα μελετήσουμε το θέμα αυτό για να καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες και θα ήθελα να συγχαρώ τις δύο συνεισηγήτρες για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γλυκόπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίζω και εγώ αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα στο σύντομο χρόνο που έχω να επικεντρωθώ σε ένα σημείο που αναφέρθηκε γρήγορα από την κυρία που ε, Είναι η ενήλικη. Και τα μεγαλύτερα θύματα είναι πραγματικά τα παιδιά και θα φροντίσουμε να κάνουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε τη θέση της προστασίας των παιδιών στην έκθεση αυτή. Η βασική τομή που θα ήθελα να φέρω είναι πρώτον. Ε, όλο αυτό το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης ε, και εισβολή στην ιδιωτική ζωή που ζούμε για αυτούς τους καιρούς είναι ιδιαίτερα δραματική για τα παιδιά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην ε, έκθεση ότι ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να το αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα το θέμα ε, της κράτησης των παιδιών ή της ακρόσης των παιδιών. Θα πρέπει να είναι χώροι που να μην αισθάνονται τα παιδιά ότι τους απειλούν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ή ας πούμε, ιατρικές εξετάσεις σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους θα πρέπει να είναι όσο γίνεται λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι και κατάλληλες ε, με την εκάστοτε περίπτωση. Και οι δικαστές θα πρέπει να σκέφτονται πάντα το συμφέρον των ε, παιδιών. Αν δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την ε, δικαιοσύνη, όπου τα παιδιά μπορεί να είναι θύματα ή μάρτυρες κάποιων αξιοπίνων πράξεων, μπορεί να μας εμπνεύσει στη δράση μας. Η ομάδα μου θα επανέλθει ε, σε αυτό το θέμα ε, της ε, αποκατάστασης δικαιοσύνη. Και ένα τελευταίο, είναι γενικότερο μάλλον σε σχέση με αυτά που είπα. Μέχρι τώρα είναι πολλές οι τροπολογίες ε, για τις αιτιολογικές σκέψεις και για κάποιες προβολές που δεν έχουν καμία νομική ισχύ, αλλά είναι διατυπωμένες με τρόπο που ε, είναι πολύ ε, βαρύγδουπος και με στόμφος, αν είχα νομική ισχύ. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τι έχει νομική ισχύ και τι όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Σέσκοβα για δύο λεπτά. Děkuji za slovo, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες, εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο και θα ήθελα να καλωσορίσω το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής που θα ενταχθεί στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα και την προστασία των θυμάτων. Έχω συνομιλήσει με εκπροσώπους διαφόρων ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, κυρίως ε, ΚΑΠΑΟ μικρών που δραστηριοποιούνται στην Τσεχία. Είμαι σίγουρη ότι χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση και ελπίζω ότι θα γίνει ακόμη σαφέστερη έκθεση και θα εγκριθεί ε, σύντομα. Θα υποστηρίξω τις τροπολογίες στο μεγαλύτερο μέρος τους, κυρίως ως προς τη δεύτερη θυματοποίηση, την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων αλλά και το μέλλον μελών της οικογένειάς τους, ε, ενημέρωση, δικαίωμα ενημέρωσης, ε, για, του, για έναν δράστη παραδείγματο χάρη που δεν κρατείται πλέον ε. σχετικά με τη βία τώρα που σχετίζεται με το φύλλο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα ούτως ή άλλως ασχολούμαι με αυτό το θέμα στην Επιτροπή των Γυναικών οι τροπολογίες 15, 16, 17 φέρουν επί ακριβώς αυτού του θέματος και θα ήθελα να τις υποστηρίξω ρητά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω μία διάσταση του ζητήματος ε, που μου σχολίασαν ε, σε πολλές περιπτώσεις οι οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία των θυμάτων. Ε, σχετίζεται λοιπόν αυτό με κάποια κέντρα υποδοχής που παρέχουν ε, υπηρεσίες προς αυτές τις κατηγορίες θυμάτων και θα ήθελα να ρωτήσω τις δύο εισηγήτριες ε, αν θα ε, υποστηρίξουν την δημιουργία τέτοιων κέντρων υποδοχών. Κύριο κύριος δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλωσορίζω τη δουλειά που κάνατε. Και πρέπει να σας πω ότι τα θύματα στην Ευρώπη έχουν τις βασικές ανάγκες. Σεβασμό, αξιοπρεπή μεταχείριση, προστασία, υποστήριξη, πρόσβαση δικαιοσύνη, αποζημίωση και επανόρθωση. Πολλά τα είπατε ήδη, ε, γι' αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω δύο ακόμα στοιχεία και να τα φέρω στο προσκήνιο. Πρώτον, ε, η πρακτική εφαρμογή ε, όλου αυτού του πακέτου. Και αυτό το συνδέω με το εξή ερώτημα. Είναι όλα τόσο ισορροπημένα ε, ώστε από πλευράς κόστους να έχουμε κάποια αναλογική ε, υλοποίηση και εφαρμογή όλων αυτών. Και μετά ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του συνόλου ε, και των δικαιωμάτων των θυμάτων που θέλουμε να αναγνωρίσουμε στα θύματα ή να τους προσδώσουμε. Μήπως αυτό παρατείνει ε, την ποινική δίωξη και τις ποινικέ δίκες και τελικά έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, στην τροπολογία 55... Τι σημαίνει επιπλέον ηλική υποστήριξη, material, Μήπως είναι έτσι γενική, πολύ γενικόλογη διατύπωση, τι εννοείται. Και στην τροπολογία 100 γίνεται λόγος για βάση δεδομένων. Μα υπάρχει ανάγκη γι' αυτό, έχουμε έτσι και λίγο στα κράτη-μέλη βάσεις τέτοιων δεδομένων. Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό για την αξιολόγηση της οδηγίας, την παρατήρηση Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκή υπόθεση αυτή γιατί η Eurostat, έχει οι εθνικέ βάσει. Η κυρία Γαρσία, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω ε, σκιώδη εισηγήτρια των σοσιαλιστών ε, στην Επιτροπή Γυναικών θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χιμένεθ Πεθερίλ και την κυρία Παρβανόβα για τη δουλειά τους. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ισχύει αυτό που έλεγε ο κύριο Ρωμέβα, ότι το θέμα αυτό δεν είναι ο μόνο χώρο στον οποίο θα πρέπει να αναφερόμαστε στα θύματα βία λόγω του φίλου τους. Εδώ και αρκετό καιρό αρκετές συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο ζητάμε μια συγκεκριμένη οδηγία για τη βία κατά ε, των γυναικών ή γενικώ ε, βία λόγω του φίλου. Βέβαια, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει ακόμα να παρουσιάσει σχετική πρόταση, θα πρέπει η οδηγία αυτή να αναφέρεται ε, συγκεκριμένα σε αυτό το κοινωνικό πλήγμα το οποίο βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι ε, κάποιοι άνθρωποι είναι θύματα απλώς και μόνο γιατί είναι γυναίκες. Ε, η βία λοιπόν λόγω του φίλου τους θα πρέπει να αναφέρεται και να έχει σημαντικό ρόλο στην οδηγία αυτή και δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή εδώ για να συζητάμε για οικονομικά ζητήματα. Όταν οι πολίτες ακούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, να γίνονται αναφορές στην οικονομική κρίση και τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα ζητήματα, το να είμαστε ε, σε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικά νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να αλλάξει ο, ε, ο τρόπος που εργαζόμαστε σε συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συγκεκριμένη μνήμα στις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει μια εγκάρσια πολιτική προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να μπορέσουμε στην οδηγία αυτή τα όλα, τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την υποστήριξη των ατόμων να ληφθούν καταλήλω υπόψη και ελπίζω να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών και των ε, συναδέλφων ανδρών και γυναικών στι δύο επιτροπέ, προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο το οποίο μα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλφάνο για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες ε, για τη δουλειά τους. Είναι πολύ περίπλοκο το έργο τους. Ιδίω όταν έχουμε ζητήματα τόσο ισχυρά και από συναισθηματική σκοπιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσουμε να καλύψουμε από νομοθετική σκοπιά τα πάντα. Ζητώ συγγνώμη, διότι δεν μπόρεσα να επισέλθω στην ουσία των προτάσεων, διότι η μετάφραση του κειμένου ε, μου ε, ήρθε χθε το απόγευμα και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Ε, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την τροπολογία 15, διότι έχουμε διάφορες κατηγορίες θυμάτων και θεωρώ ότι μπορώ να είμαι ευτυχής ε, διότι στις κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματο. Με ενδιαφέρει επίσης ε, το θέμα του δικαιώματο στην προστασία, της ασφάλειας, ε, του δικαιώματος να γνωρίζει κάποιο την αλήθεια και να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη κάποιων γεγονότων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλέ φορέ λησμονούνται και μένουν στο από της ιστορίας κάποια θέματα. Τερέζα και Αντώνια δεν θα συνεισφέρω μόνο ως βουλευτής αλλά και ως πρόεδρος της ε, ε, ε, οργάνωσης που έχουμε στην Ιταλία για τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας. Και εσείς έχετε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι των ατόμων που ε, είναι θύματα και τα μέλη της οικογένειας θυμάτων και το καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντάξουμε ε, στα θέματα των θυμάτων και θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τα μέλη της οικογένειας θυμάτων στα θύματα. Θα σας κάνω και σχετική πρόταση τροπολογίας. Ο κύριος Μπρόνς για δύο λεπτά. It's not responding, right. The rights of victims of crime τα δικαιώματα των θυμάτων είναι αυτονόητο ότι είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε και ποιε είναι οι επιπτώσει των εγκληματικών πράξεων σε συγκεκριμένα πλαίσια, σε συγκεκριμένε κοινωνίε. Ε, δεν ε, θεωρώ ότι συντρέχει λόγο να συνιστά αυτό προτε... Ε, αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Επίση, ε, υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου δεν καλύπτονται τα δικαιώματα των θυμάτων σε κάποιες κοινωνίε. Μα έλεγε η Δανική Προεδρία σήμερα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να νομοθετούν. Μα ήδη την έχουν. Και μάλιστα έχουν εγκρίνει πολύ αποτελεσματικά νομοθετήματα, κάποια από αυτά. Ε, δεν νομίζω ότι είναι ο σκοπό η εναρμόνιση της ε, νομοθεσίας, είτε μιλάμε για το Κοινοβούλιο είτε για τα κράτη-μέλη. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση και να χαρακτηρίζουμε ως ευάλωτα κάποια θύματα. Ε, στην, ε, στο αγγλικό κείμενο στη σελίδα 63 δείτε πόσο αποκαλυπτική είναι η διατύπωση. Και λέει, αλλά σβήνει το μικρόφωνο του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 Φαίνεται ότι η κινητήριο δύναμη των νομοθετών ε, ε, εδώ όπω και αλλού είναι να ανάγουν σε αυτό σκοπό την εναρμόνιση τη νομοθεσία. Ε, και όταν μιλάμε για βασικέ αρχέ όπω διεθνή κινητικότητα των ανθρώπων και κατάργηση τη διακριτική μεταχείριση, αυτοί εστιάζουν μόνο στα θύματα. Δείτε στην τέταρτη παράγραφο, σελίδα 63 του κειμένου, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, λέει εδώ ότι η αναγνώριση της βίας κατά των γυναικών είναι μορφή διακριτικής μεταχείρισης ε, που πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοια και να καταπολεμηθεί. Όλοι καταδικάζουν τη βία εναντίον των γυναικών, αλλά αυτό, αυτή η διατύπωση δίνει την εντύπωση ότι ε, η βία που συνδέεται με το φύλλο ε, θεωρείται ως ε, διακριτική μεταχείριση και αυτό είναι πιο σημαντικό από την ίδια τη βία. Νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο για δύο λεπτά παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Η οδηγία του Συμβουλίου αν την εξετάσουμε από την οπτική του κράτους δικαίου δεν εισαγάγει τίποτα, διότι υπάρχουν τα δικαιώματα των θυμάτων στις ε, δικαστικές διαδικασίες. Βεβαίως, ε, το γεγονός ότι υπάρχει μια οδηγία σημαίνει ότι το Συμβούλιο νιώθει την ανάγκη να τυποποιήσει κατά κάποιο τρόπο και να ομογενοποιήσει μεταξύ των 27 κρατών μελών ε, πράγματα τα οποία είναι ακόμα και τα συνήθι δικαιώματα που έχουμε στο κράτος δικαίου. Δεν βλέπω και καμιά επανάσταση σε αυτή την έκθεση. Οι δύο εισηγήτριες έχουν κάνει κάποιες ε, σημαντικές καινοτομίες όσον αφορά την προάσπιση των μειονοτήτων. πολύ σημαντικά κίνητρα και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ε, επέστησαν την προσοχή μας ε, στα θέματα των μειονοτήτων ή αν θέλετε ε, όχι μειονότητες, άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα φύλου, τα προβλήματα των παιδιών, τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες ή αναπηρίες. Διερωτώ με όμως, η ανάγκη να προασπίσουμε που αντιμετωπίζουν, αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, όχι μόνο στις δικαστικές διαδικασίες, αλλά ακόμα και στην ίδια την κοινωνία, για λόγους προκαταλήψεων, ρατσισμού, ή και λόγω της ε, ε ταυτότητας του φίλου τους ε, αφορούν μόνο τις γυναίκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Μία μαύρη γυναίκα είναι μάλλον αντικείμενο περισσότερη διάκριση από ότι μια λευκή γυναίκα. Οι μετανάστες έχουν ή δεν έχουν το δικαίωμα συγκεκριμένη αναγνώριση στις δικαστικές διαδικασίες και οι μειονότητες. Θα ήθελα να αναφερθώ σαφέστατα στην νομοθεσία που έχουν διάφορες χώρες για τους ομοφιλόφιλους, ε, τους ε, ε, αμφιφιλόφιλους και ούτε καθεξής. Τι γίνεται, τους τα δίνουμε αυτά τα δικαιώματα ή πρόκειται για δικαιώματα τα οποία εστερνιζόμαστε σε γενικές γραμμές αλλά δεν εφαρμόζουμε σε πολλές περιπτώσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και σε πολλά άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη δεν αναφερόμαστε σε συλλογικά εγκλήματα, πράξεις τρομοκρατίας, ε, πράξεις ε, οι οποίες καταστρέφουν το περιβάλλον. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει σαφέστατα στην έκθεση αυτή να αναφέρει τη δυνατότητα της συλλογική προσφυγής, δηλαδή της συλλογική αγωγής, ε, δυνατότητα οργανωμένες ομάδες μειονοτήτων που έχουν υποστεί ζημίες ή έχουν ε, υπάρξει θύματα να μπορούν να καταθέσουν αγωγή συλλογικά και να βρουν ε, το δίκιο τους. Ε, κύριε Κροτσέτα, είμαι βέβαιο ότι όταν αναφερθήκατε στη σύγκριση μεταξύ μιας μαύρης και μιας συνηθισμένη γυναίκας, δεν θέλετε να πείτε ότι μια μαύρη γυναίκα δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα. ίσα ίσα, ίσω πιο συνηθισμένη από τι υπόλοιπε, απλώ λέω ότι στη σημερινή κοινωνία είναι αντικείμενο διπλή διάκριση και για το χρώμα του δέρματός τη, αλλά και για το φύλλο τη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει η διευκρίνηση. Η κυρία Κλάς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ερώτηση έχω εγώ στην εισηγήτρια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ορισμό του θύματος εγώ έτσι όπως το κατανοώ, είναι θύματα μιας αξιόπινης πράξης. Τι γίνεται όμως με τα θύματα ε, των ε, υπευθύνων, των ενόχων, δηλαδή γενικότερα όχι μόνο της πράξης και η οικογένεια, τα παιδιά κάποιου, ας πούμε. Δεν είναι και αυτοί θύματα, δηλαδή οι συγγενείς ε, του ε, ενόχου, ο οποίος έχει καταδικαστεί και κρατείται στη φυλακή. Έχουμε καθυστερήσει, λέει ο Πρόεδρος, το έχετε διαπιστώσει κι εσείς άλλωστε. Προσπαθώ να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο έκαστος. Αλλά βλέπετε ότι όλοι μίλησαν τρία λεπτά και καθυστερήσαμε. Έχουμε όμως και ψηφοφορία στις 10 και 4 προγραμματισμένη και πάντα την ίδια ιστορία ζούμε. Ορισμένοι έχουν προγραμματίσει να έρθουν μόνο στη ψηφοφορία στις 10 και 4 και έρχονται γι' αυτό. Λοιπόν, αν θέλουν οι συγγήτριες ένα λεπτό η κάθε μία να ολοκληρώσουν, να ευχαριστήσουν ξέρω εγώ τι θέλετε και μετά να περάσουμε στο επόμενο θέμα για να προκάνουμε διαδικαστικό, κύριο Μπουσουτήλ. Ναι, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψηφοφορία πάση θυσία να γίνει εγκαίρω. Διότι ορισμένοι ακριβώ έρχονται ακριβώ για την ψηφοφορία και μετά φεύγουν. Ακριβώ αυτό είπα κι εγώ, λέει ο Πρόεδρο. Συμφωνώ 100%. Eh. Κυρία Χιμένε Πεσερίλ, Ακριβώ επειδή δεν έχουμε χρόνο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ρωτήσατε και είπατε. Ε, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, δεν θα το κάνω τώρα, διμερώς ή αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, θα τα συζητήσουμε αυτά και θα φροντίσουμε και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέσφεραν. Η κυρία Παρβάνοβα, ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και τις τροπολογίες. Όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη με μεγάλη προσοχή. Θέλω μόνο να πω σε ό,τι αφορά τη βία με βάση το φύλλο, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Δεσμεύτηκε προσωπικά η κυρία Ρέντινγκ, η Επιτροπός ήδη κατά τη διάρκεια της ακρόασης της και μετά σε συνεδριάσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι αυτή είναι η ευκαιρία, αυτή είναι η κατάλληλη θέση να μιλήσουμε για βία ε, με βάση το φύλλο. Και αυτό συνάδει πλήρως και συμμορφώνεται με την προστασία των γυναικών ε, κατά τα άλλα αυτό το έχουν κυρώσει όλα τα κρατημέλη και έχει δεσμευτική ισχύ, ξέρετε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Πρόεδρος, τώρα, κοιτάξτε τι έχουμε. Έχουμε το σημείο 4 για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, του 2013. Και είναι και η κυρία Παπαδοπούλου παρούσα εισηγήτρια. Το θέμα όμως είναι ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 10 και 4. Εάν θέλετε όμως, κυρία Παπαδοπούλου, να κάνετε εσείς την παρουσίασή σας και μετά να ψηφίσουμε. Για να αρχίσουμε στις 10 και 4 ακριβώ ψηφοφορίες. Συμφωνείτε, κυρία Παπαδοπούλου. Yes. I will have to... Ευχαριστώ. Και εγώ έχω αεροπλάνο να προλάβω, οπότε πρέπει να παρουσιάσω τώρα την ε, πρόταση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη, ε, ούτω ώστε να γίνει Ευρωπαϊκό Έτο των Πολιτών το 2013. Πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλο, ε, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Έτο θα πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Έτο τη Ιθαγένεια και όχι των πολιτών, ε, όπω είπε το Κοινοβούλιο 15 Δεκεμβρίου 2010 στο σχετικό ψήφισμά του, διότι μιλάμε τα... και επίση στο ψήφισμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε άλλο ψήφισμα το 2009. Έτσι μπορούμε να αυξήσουμε την ενημέρωση των πολιτών για την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια, να τονώσουμε ε, την ε, συμμετοχή τους στα κοινά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εμπόδια και δημοκρατικά ελλείμματα και τα μεγάλα ποσοστά αποχής στις ευρωπαϊκές εκλογές. το 83, όπως ξέρετε, το 93 μάλλον η συνδίκη του Μάστριχτ προέβλεψε για πρώτη φορά την ηθαγένεια και τώρα... Μετά από τόσα χρόνια, οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ θόρυβο μέσα στην αίθουσα. Δεν μπορώ να παρουσιάσω στην την έκθεσή μου. Please, dear colleagues and members. Αγαπητοί συνάδελφοι. So, please, let's pay attention to πρέπει να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση. Σας παρακαλώ να προσέξετε, αυτή, να δώσετε βάση στην παρουσίαση. Ας αφήσουμε την κυρία Παπαδοπούλη να κάνει την παρουσίαση της. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απολάβουν πάρα πολλών δικαιωμάτων, όχι μόνο την ελευθερία της ε, την κινητικότητα που έχουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να είναι υποψήφοι σε ευρωπαϊκές εκλογές και να ψηφίζουν στη χώρα που διαμένουν, να έχουν ε, προστασία από τις διπλωματικές και φιλοξενικές αρχές ε, μπορούν ε, να υποβάλουν έτοιμα στον Ευρωπαϊκό ε, Διαμεσολαβητή, μπορούν να αποταθούν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες. Λοιπόν, πιστεύουμε για αυτούς τους λόγους ότι αυτό το ευρωπαϊκό έτος της Ιθαγένειας θα πρέπει να τονώσει το, τις γνώσεις των πολιτών σε σχέση με όλα αυτά τα δικαιώματα όπου και αν διαμένουν μέσα στην Ένωση. Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις μετα μεταξύ των οποίων αναγνωρίζουμε την ανάγκη συμμετοχής στα κοινά των πολιτών της Ένωσης, την ανάγκη καταπολέμησης, ε, όπως έλεγα, του δημοκρατικού ελλείμματος και του υψηλού ποσοστού αποχής στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα διοργανώσουμε εκστρατείες ε, ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ε, θα προβάλλουμε αυτό το ευρωπαϊκό έτος στα ΜΜΕ και άλλο. Προτείνουμε σχέδιο δράσης και συγκρότηση μιας ειδικής καθοδηγητικής επιτροπής και μιας task force για την Ιθαγέννη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προτείνουμε πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την ηθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 καθώς και έγκριση πράσινη βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να δρομολογήσουμε ολοκληρωμένο διάλογο για την ενεργό ηθαγένεια. Επιπροσθέτως, αυτό το θέμα του συγκριτικού εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου διευκρινίζονται ε, οι όροι έχει καθοριστική σημασία. Ένα εκατομμύριο ευρώ είναι το κονδύλι για φέτος. Αν ε, κάνουμε μία σύγκριση με χρηματοδότηση προηγουμένων ετών θα διαπιστώσουμε πόσο πενιχρά είναι τα κονδύλια. Το 2011 ε, είχαμε ένα κονδύλι 11 εκατομμυρίων για την εκστρατεία και το 2012 2010 27 ε, εκατομμύρια. Φέτος το 2000 για το 2013 μάλλον προβλέπεται μόνο ένα εκατομμύριο. Φυσικά δεν επαρκεί διότι δεν προβλέπεται καμία συγχρηματοδότηση για πρωτοβουλίες ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, και οργανώσεων των πολιτών ούτως, ούτως ώστε να εφαρμοστούν τα κατάλληλα επικοινωνιακά μέτρα για την ενημέρωση. Προτείνουμε λοιπόν αύξηση του κονδυλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος προτείνουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος της Ιθαγένειας να μην είναι μια απλή επέτειος, να προσπαθήσουμε να γίνει η αρχή συγκρότησης ενός πλαισίου ε, για μακροπρόθεσμο διάλογο για αυτήν την ε, ενεξελίξη έννοια της Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε οδικό χάρτη που θα λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικέ πολιτικές, ε, μελλοντικά σχέδια και δράσεις που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αναμένω τροπολογίες των συναδέλφων ο στόχος του έτους είναι να βελτιωθεί η κατανόηση από πλευρά των πολιτών της ευρωπαϊκής ιστορίας και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παπαδοπούλου, που ήσασταν τόσο σύντομοι. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε ένα πρόβλημα, όπως έλεγα. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα στις και τέταρτο την ψηφοφορία. Ταυτόχρονα εξετάζουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ο κύριος Σόγκορ θέλει το λόγο. Παρακαλώ, αν θέλετε το λόγο για ένα-δύο λεπτάκια, αλλά μην τα υπερβείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα τα πω ουγγρικά. Ναι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη εισηγητής του Λαϊκού Κόμματος και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός καν ότι έχουμε μια τέτοια έκθεση. Η Ευρώπη δεν διανύει μόνο οικονομική κρίση, αλλά και ηθική, πρέπει να σας πω. Συχνά Μας υβρίζουν, μας προσβάλλουν, μας επικρίνουν, μας λιδωρούν οι πολίτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε μια τέτοια συζήτηση. Πρόκειται για την κοινωνική προστασία. Ξέρουμε τι προβλήματα έχουμε όλοι με την κοινωνική μας προστασία. Ε, τα συστήματα πρόνοια, τα πανεπιστημιακά διπλώματα, δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντικό. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε σύντομοι, κυρία Γκρισμπέκ. Έχετε το λόγο, αλλά για πολύ λίγο. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Συρρυκνώνεται συνεχώς ο χρόνος που μας δίδεται. Για την έκθεση αυτή θέλω να τονίσω την πάρα πολύ υψηλή ποιότητα της εργασίας ε, της εισηγήτριας συναδέλφου μας, η κυρία Αντιγόνης Παπαδοπούλου. Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Δεν γεννιέσαι πολίτης, γίνεσαι. Και δεν είναι κατάσταση, είναι μόνιμη και διαρκής κατάκτηση το να είσαι πολίτης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση πίσω από την έκθεση αυτή που μπορεί να φαίνεται ε, αξιοπερίεργη γιατί υπάρχει κρίση και δυσκολίες αλλά ο χαρακτήρας του Ευρωπαίου πολίτη και η ηθαγένεια απομακρύνεται συνεχώς από τους Ευρωπαίους πολίτες. Λοιπόν, είτε θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη ή η έννοια τη Ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια ε, είναι τεράστια, εξαπλώνεται πάρα πολύ, δεν είναι περιοριστική όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ συμφωνώ με την εισηγήτρια. Δεν είναι απλώ ένα νομικό καθεστώ ελεύθερη κυκλοφορία και τελείωσε. Θα πρέπει να έχουμε και ένα όραμα ε, ευρύτατο τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια σε όλου του τομεί εγκάρσιο και με την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κυρία Τζάνοκα, σύντομα παρακαλώ. Τελευταία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρέπει να πω ότι ε, συμφωνώ να αλλάξει ο τίτλος, να μιλάμε για ηθαγένεια και όχι για πολίτες. Είναι ευρωπαϊκό έτος ηθαγένειας. Θα πρέπει να το συζητήσουμε να αλλάξει. Ευρωπαϊκό έτος ηθαγένειας, όχι ευρωπαϊκό έτος των πολιτών. Θα έχουμε και άλλες συζητήσεις. Ε, υποστηρίζω πλήρως κυρία Παπαδοπούλου σε αυτό το θέμα και θα, εν ευθέτω χρόνο θα μπούμε και σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και θα πούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα, περίπου στην ώρα της, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, να σας πω, πριν τελειώσουμε αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ, προσέξτε με λίγο. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία για να ψηφίσουμε. Θυμίζω, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση της κυρίας Παπαδοπούλου έχει οριστεί 21 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Τροπολογίες. 21 Φεβρουαρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι ακριβώς. Ωραία. Προχωρούμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έχουμε προγραμματίσει. Και επειδή έχω κάτι θεσμικά που δεν μπορώ να αποφύγω, θα παρακαλήσω την κυρία Κίνγκα Γκόνς να αναλάβει την Προεδρία για την επόμενη ώρα, γιατί είμαι αναγκασμένος να φύγω. Και ψηφίζουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Μόλις έμαθα ότι έπρεπε να προεδρεύσω. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ευνηδιάζουμε έτσι τον κόσμο στην Επιτροπή μας. The first, uh, vote on... Uh, Η πρώτη ψηφοφορία λοιπόν στη μερίσια διάταξή μας είναι έκθεση 210 για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια ήταν η κυρία Σδανόκα. Ποια στιγμή να βγάλω τη γάρτα μου για να ψηφίσω. Η συμβαστική υπαριθμών 1. Ψηφί Κατά. Αποχές. Α, εδώ χρειάζεται έλεγχος. Παρακαλώ, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. I open the vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Αλλάξτε θέση όσοι δεν ε, ε, έχετε μηχανήματα που λειτουργούν και θα προσθέσουμε το όνομα τας. Ωραία, λειτουργούν όλα. Πέρες. 26 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Οι 4 καταπίπτει και μερικές άλλες ακόμα. Και πάμε στη συμβαστική υπαριθμό 2. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική υπαριθμό 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Τι θέλετε, έλεγχο για τη συμβαστική 4 της αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. 24 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 10. Ψηφί πε. Κατά. Αποχές. Πολύ δύσκολο να καταλάβω. Δεν σηκώνεται και χέρια. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την τροπολογία υπαριθμών 10. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 10. Απερίφθη η συμβιβαστική, γι' αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες. Και τώρα είμαστε στη 10. Πέρας. Okay, now I close Πέρας. 16 υπέρ, 38 κατά, απορρίπτεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω. Ε, χρειάζεται έλεγχος. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Now we close the vote. Πέρασε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μου λέει γραμματεία περισσεύει ένας. Είστε υπεράριθμοι. Τώρα εντάξει. Βγάλετε μια κάρτα. Εντάξει. Πέρας. Μόνο για αυτή την τροπολογία ήταν, δεν ήταν τη συμβαστική. Τα παρακολουθεί η γραμματεία αυτά. Πέρας. 26 υπέρ, 27 κατά. Καταπίπτει. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πάλι ηλεκτρονική υπαλήθευση χρειάζεται. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία 26-26 απορρίπτεται. Έχει συμβιβαστική παριθμό 5. ψηφιπέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στη συμβαστική παρελθόν 6. Ψήφι κατά αποχέ. πάλι χρειάζεται έλεγχος τα ίδια. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελειώνει. ισοψηφία και πάλι απορρίπτεται. Η τροπολογία 20 ψήφι Κατά. Αποχές. Rejected. 21. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. αυτό τώρα τι είναι. Έλεγχο θέλει. Ζητώ συγγνώμη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για την 21. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Πέρασε. 25 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην 24. Ψήφι Κατά. Αποχές. Έλεγχος και πάλι χρειάζεται. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας το λέξουμε. Πέρασε. Πέρας. ψηφιο ισοψηφία 26-26 απορρίπτεται. Και μία αποχή πάντα. 25 και 26 μαζί, γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές και πάλι έλεγχος. Οι ίδιες ε, ιστορίες πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. in favor, 27 against, 1... 24 υπέρ, 27 κατά, μία αποχή, απορρίπτεται. 23 υπέρ. Against. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική υπαριθμόν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική, όχι, μισό λεπτό. Ναι, η συμβαστική 10. Υπέρ, κατά. Συμβιβαστική υπερθμόν 10 και θα χρειαστεί έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε σας παρακαλώ πολύ. Πέρασε. Πάλι παρσεύει ένας από το ΕΛΚ. Βγάλετε παρακαλώ κάποια κάρτα. Ξαναψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 29 υπέρ, 22 κατά. Δύο εποχές. Εγκρίνεται. Η συμβιβαστική υπαριθμόν 11 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. I open the vote. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. 27 υπέρ 24 ε, κατά, δύο εποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στη συμβαστική 12 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise Amendment 14 in favor. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise amendment. Η συμβαστική 15 είπε κατά αποχές νομίζω ότι είχε απορριφθεί αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. The vote is closed. 26... Πέρασε 26 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. Μάλιστα. So we have to vote on 62, 63, 64. 62, 63, 64 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 27 in υπέρ, 26 κατά χωρίς αποχές συγκρίνονται. Αυτές οι τρεις. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία... Όχι, δεν ερχόμαστε, καταπίπτουν. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε το σύνολό του. Όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν. Πάμε στην τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Α, όχι, εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μου είχε διαφύγει. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ακόμα ψηφίζουμε. Δεν έχετε ψηφίσει όλοι ακόμα. Πέρες. 25 υπέρ, 25 κατά και δύο εποχές. Απορρίπτεται το σύνολο της νομοδότησης. The next vote. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Απαλλαγή 2010, Γενικός Προϋπολογισμός, τμήμα 3. Συντάκτης ο κύριος Βαντεκάμπ. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία. Επομένως άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης υπέρ, κατά, αποχές. Συγγνώμη, έχουμε μόνο την τελική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικός, λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Σχέδιο γνωμοδότησης για το τμήμα 3 της Επιτροπής. Πέραση της ψηφοφορίας. 49 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Κατόπιν, Σχέδιο γνωμοδότησης απαλλαγή 2010, Γενικό προπολογισμό, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Και πάλι μόνο μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρασε ψηφοφορία. 50 in 50 υπέρ, κανείς κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Απαλλαγή 2010, απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι μία ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. close the vote. 48 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Ε, draft opinion. Γνωμοδότηση για την απαλλαγή Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010. Τρεις τροπολογίες. Υπέρ της πρώτης, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς για το σχέδιο της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. Πέρασε της ψηφοφορίας. 50 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται και τώρα ε, γνωμοδότηση για τα εξωτερικά σύνορα ε, των κρατών μελών, η Frontex, 7 τροπολογίες, πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο στροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρασε ψηφοφορίας. Συγγνώμη, έγινε κάποιο λάθος. Πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Please vote. Ψηφίστε παρακαλώ. I close the vote. Πέρασε η ψηφοφορία. 49 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μπουσουτήλ. Προχωρούμε. Απαλογή της Europol για το 2010. Μία τροπολογία εδώ, υπέρ της τροπολογίας 1, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο σου τροποποιήθηκε, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. ψηφοφορία. 50, in favor. 50 μία κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Κατόπιν. Δεύτερη γνωμοδότηση της κυρίας Σόμερ. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. ψηφοφορίας. 49 ψήφοι υπέρ, κανείς κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ζόμερ. Περνάμε τώρα στην απαλλαγή 2010 για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Η συντάκτρια είναι η κυρία Ματιέ. Τέσσερις τροπολογίες. Πρώτη, υπέρ. Who is against? Κατά. Αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote, please, colleagues, vote, because it's... Παρακαλώ ψηφίστε συνάδελφοι. Okay. I close the vote. Πέρασε της ψηφοφορίας. 19 ψήφοι υπέρ, 31 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ψηφο. close the vote. Πέρασε τη ψηφοφορία. 48 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κυρία Ματιέ. Γνωμοδότηση για την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Παρατηρήτητο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το 2010. Ε, συντάκτης ο κύριος Ιακολίνου. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. We can close the vote now. Πέραση ψηφοφορία. 44 ψήφοι υπέρ, Κανεί κατά, τρει αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κυρία Κολίνο. Okay. As I was informed, there was a... Uh, όπως με ενημέρωσαν, είχε προβλεφτεί και μια ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Κοέλιο, αλλά αναβλήθηκε και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένετε μισό λεπτό. I ask you colleagues to leave the room. Συνάδελφοι, παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να εξηγήσω κάτι στους συναδέλφους. Why I'm asking for the postponing of... Ζητώ αναβολή ε, της ε, ψηφοφορίας. Κύριε Κοέλιο, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, πρέπει να αποχωρήσετε αν θέλετε να συζητήσετε με τους συναδέλφους. Continue this way. Thank you. Thank you, Mr. Thank you so much. Uh, I was uh, explaining... Ε, ο κύριος Κοέλιο, πρόεδρε, θέλω να εξηγήσω γιατί ζήτησα μετάθεση της ψηφοφορίας. Ε, οι συνάδελφοι έχουν λάβει την επιστολή της Δανικής Προεδρίας ε, όπου ζητείται έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο για το περιεχόμενο της πρότασης δεν νομίζω ότι πρέπει να αρνηθούμε αυτή την πρόσκληση προς ε, διάλογο. Δεν θα ψηφίσουμε την αλλαγή ε, της ε, νομικής βάσης. Το Συμβούλιο δηλαδή δεν πρόκειται να ξεκινήσει πόλεμο, αν θέλετε, κατά του Κοινοβουλίου. Πρέπει να απαντήσουμε θετικά. Πρέπει να δεχτούμε την έναρξη του διαλόγου. Θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία ή στη Λίμπε ή στην Ολομέλη. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διατάξεως, δηλαδή το υπαριθμόν 16. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2008 έως 2013. Uh, ε, as you remember, the θα θυμάστε ότι το θέμα της μετεγκατάστασης, της αποκατάστασης των προσφύγων είχε παγώσει στο Συμβούλιο. Στο μεταξύ στις 18 Μαΐου 2010 εγκρίθηκε η θέση για την πρώτη ανάγνωση. Μετά επανήλθε το Δεκέμβριο του 2010 το θέμα στο Συμβούλιο και η Ιδανική Προεδρία έχει εντολή για να διαπραγματευτεί την ε, κοινή θέση του Συμβουλίου της πρώτης ανάγνωσης έχει ε, κατανεμηθεί αντίτυπο σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή. Θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μα, τον κύριο Ταβάρε. Είναι εδώ ο κύριο Ταβάρε. As... We don't see the rapporteur. Δεν βλέπω τον εισηγητή. So, uh, we should give the floor to the Άρα θα δώσουμε το λόγο στο Συμβούλιο τότε. Αφού δεν έχει καταφτάσει ο εισηγητής, ε, θα δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή, μετά στο Συμβούλιο και μετά επιστρέψουμε στον εισηγητή μας. Ε, παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε εκείνος είναι. Πολύ ωραίο. Is here from the Είναι κανείς εδώ που να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Έχουμε, έχουμε εκπρόσωπο, αλλά θέλουμε να ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή πριν τοποθετηθούμε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά εν τη αυτή περίπτωση θα περιμένουμε, ξέρω εγώ, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, μονόλεπτο. One minute, because it's supposed to start at έχει προγραμματιστεί για τις 11 παρατέταρτο το σημείο αυτό. Ας περιμένουμε αυτό το λεπτό που υπολείπεται. I heard that the reporter is... Μου σφύριξαν ότι έρχεται ο εισηγητή, είναι σε άλλη επιτροπή. For us to be present at two places at one time. Ο εκτός αν κλωνοποιηθεί να είναι σε δύο επιτροπές ταυτόχρονα. for the rapporteur. Okay. I think we can continue. Μάλιστα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Καλώς ορίσατε κύριε Ταβάς. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο μετά την εισαγωγή μου. Μετά θα ακούσετε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρακαλώ κύριε Ταβάρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί αργοπόρησα ελαφρώς, αλλά ήμουν Δύο ρόφου παραπάνω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συζητούμε τι στρατηγικέ επιπτώσει ε, τη αναθεώρηση πολιτική περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπήρξε μια μικρή σύγκρουση. Είναι και τα δύο θέματα τέλος πάντων ε, σημαντικά και θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι ο φάκελο συναπόφαση ε, σχετικά με του κανόνε που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων είναι κάτι που μα απασχολεί από τα τέλη του 2009 και έχουμε εγκρίνει ήδη το Μάιο του 2010 την ε, έκθεση. Ταυτόχρονα την έκθεση συναπόφαση. Ταυτόχρονα εγκρίναμε το ψήφισμά μα ε, σχετικά με την μετεγκατάσταση και αποκατάσταση των προσφύγων Έχει εργαστεί σκληρά το Κοινοβούλιο, υπήρξε ομοθυμία σε σχέση με εκθέσεις και ψηφίσματα στο, για το ίδιο θέμα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φάκελο. Είναι άνθρωποι που είναι σε καταβλισμούς προσφύγων, ε, διαβίουν σε καταβλισμούς προσφύγων και έχουν ε, διατρέξει κίνδυνο για τη ζωή τους ακόμη πριν φτάσουν στον καταβλισμό. Εγκαίρως λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε το νομοθετικό κομμάτι για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Δυστυχώς ε, ε, υπήρξαν πολλά εμπόδια καθοδόν ε, οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση, τα εφαρμοστικά μέτρα είναι θέματα που μας απασχόλησαν επί μακρό και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν καταφέραμε ε, να επιτύχουμε κάποια κινητοποίηση, δράση του Συμβουλίου. Έκανε κάποια κίνηση στο Συμβούλιο πρόσφατα. Χαίρομαι για τη συνεργασία με την ε, Δανική Προεδρία. Έχει σημειωθεί πρόοδος χάρη σε αυτή τη συνεργασία. Οι σκιώδεις ε, των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων γνωρίζουν ότι χρειάστηκε να είμαστε και ε, ευρηματικοί ε, ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Έπρεπε να βρούμε αντικατάστατο για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Έγινε αυτό τελικά σε συζητήσεις με την Ουγγρική Προεδρία, διότι εκείνοι υπέβαλαν μια σχετική πρόταση. Εμείς καταθέσαμε αντιπρόταση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να ρυθμιστεί το πρόβλημα με αυτές τις προτάσεις. Τώρα έχουμε νέα πρόταση από πλευρά της Δανικής Προεδρίας. Αυτή η πρόταση, κατά τη γνώμη μου, καλύπτει πλήρως την, ε, το διτό ε, χαρακτήρα της ε, πολιτικής μας ε, που θέλουμε να καλύπτει το νέο νομοθέτημα. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων πρέπει πρώτα απ' όλα να εξυπηρετεί ανθρωπιστικούς σκοπούς και άρα να χρησιμοποιείται για να βοηθούμε τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες. Το Κοινοβούλιο προέκρινε το σαφή προσδιορισμό ε, επιμέρους ε, κατηγοριών ε, λί ανεβάλλοντων προσφύγων που πρέπει να προστατευτούν και δέχτηκε αυτήν την ταξινόμηση στο Συμβούλιο πάρα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη όμως αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο είναι επίσης ένα πολιτικό εργαλείο και είναι σημαντικό να ενταχθεί στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των κρίσεων, για την ε, δράση μας στον τομέα αυτό και εξυπηρετεί και στόχους εξωτερικής πολιτικής. Για να δράσει με στρατηγικά λογικό τρόπο για την αποκατάσταση των προσφύγων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στους πλέον κέριους τομείς να έχει εστιασμένη δράση και να επικεντρώσει τη δράση της σε στρατηγικές περιοχές δράσης. Αυτό συνεπάγεται ότι επανειεραρχούνται οι προτεραιότητες αλλά είναι απαραίτητο. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση για τις περιφερειακές προτεραιότητες, διότι το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα ε, της διατηρεί τις προτάσεις μας στη θέση του το Συμβούλιο έχει και ένα παράρτημα με περιφέρειες προτεραιότητας ε, πέραν των προγραμμάτων προτεραιότητας ε, που ήδη τρέχουν οι πιο σημαντικοί περιοχές ε, του κόσμου, δηλαδή όπου χρειάζεται ε, κατεπηγόντως και έχει ιδιαίτερη σημασία η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έγγραφο του Συμβουλίου βλέπουμε τρεις ε, βασικές ανησυχίες ε, που συζήτησα ήδη με τους ε, σκιώδεις συζητητές και έχουμε γύρει αυτά τα ζητήματα στις κοινέ συνεδρίες με άλλες πολιτικές ομάδες. Τρία συν ένα, έτσι, τρία, τρεις βασικές ανησυχίες συν μία. Ας αρχίσω με τις βασικές ανησυχίες. Στις ανθρωπιστικές κατηγορίες. Ε, στην πρώτη διαδικασία στην απόφαση το Κοινοβούλιο είχε εισαγάγει μια νέα κατηγορία που έχει ύψιστη προτεραιότητα για μας. Ε, δηλαδή όσοι έχουν επιβιώσει ενώ έχει ασκηθεί βία ή έχουν υποστεί ε, βασανιστήρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για ανθρωπιστικούς λόγους. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στον επερχόμενο τριμερή διάλογο. on the regional... Σχετικά τώρα με τις περιφερειακές προτεραιότητες, ε, μάλλον τις προτεραιότητες ως προς τις περιοχές του κόσμου, που πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα, όλες αυτές οι περιοχές είναι στον αντίστοιχο κατάλογο του, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Οι, προ... οι Ιρακινοί πρόσφυγες είναι μεταξύ αυτών των ε, ε, περιοχών προτεραιότητας ε, και στη συζήτηση που είχαμε με τους Σκιώδης θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για τους πρόσφυγες που προέρχονται από το Ιράκ, όχι μόνο για τους Ιρακινούς, διότι υπάρχουν μειονότητες Παλαιστίνοι, παραδείγματο χάρη, που ζουν στο Ιράκ και έχουν υποστεί ε, θρησκευτικούς και άλλους διωγμούς. Πρόκειται και για χριστιανούς και για μουσουλμάνους Φέρει Φερρυπίν ε, στη Συρία σε ένα καταβλισμό προσφύγων επειδή έγινε επίσκεψη από το Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει κλείσει ο καταβλισμός από το 2010 παραμένει ανοιχτός ε, ε, είναι μεγάλος αριθμός των προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν λέμε πρόσφυγες από το Ιράκ να εννοούμε όχι Ιρακινούς, Ιρακινείς γίνει, αλλά γενικότερα πρόσφυγες που προέρχονται από τη χώρα Ιράκ και άλλων εθνικότητων Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έγιναν κάποιες πολιτικές ομάδες, σε όλες ιδιαίτερα στο ΕΛΚ, είναι το εξής. Ε, τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας ε, που καλύπτουν τις μεγάλες λίμνες, ε, την Τανζανία, την Ανατολική Ευρώπη, την Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, το κέρας της Αφρικής, Τζιμπουτή, Κένια, Ιεμένη, Βόρεια Αφρική, Αιγυπτή το Σολιβίμ, την Ισία, ε, Σχάτος. Επισκεφτήκαμε και εκεί καταβλισμούς προσφύγων, συγκεκριμένα τον καταβλισμό Σούσα που συζητήσαμε πριν από δύο ημέρες. Ε, αυτά τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας ή μάλλον αυτές οι περιοχές που καλύπτονται πρέπει να ε, προβληθούν μέσα ε, στο τελευταίο κείμενο και όπως σας έλεγα έχουμε τρεις συν μία ανησυχίες, τρία συν ένα προβλήματα. Αυτή είναι η τρίτη λοιπόν ανησυχία που έχουμε ε, και είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όπως σας είπα, στον επερχόμενο τριμερή διάλογο. Τρεις συν μία ανησυχίες είπα στις απαρχές της διαδικασίας Είχαμε ένα πρόβλημα μάλλον τεχνικής και όχι τόσο πολιτικής φύσης. Ε, το θέμα της νομικής βάσης. Βασιστήκαμε σε δύο άρθρα της συνθήκης, το 79-6G, ε, σχετικά με την ε, κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση μεταναστευτικών ε, ροών και εκπώνηση κοινή πολιτικής ασύλου και άρθρο 80 αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτά τα δύο συνιστούν τη νομική βάση. Ε, στο, στην κοινή θέση του Συμβουλίου όμως ε, δεν προβλέπεται το άρθρο 80 ως νομική βάση πλην όμως ε, το Κοινοβούλιο πρεσβεύει πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ε, πρέπει να βασίζεται σε αυτό το άρθρο για την αλληλεγγύη όχι μόνο προς τους πρόσφυγες αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως προς τη διαχείριση ε, τη αυτή περιπτώσει του προγράμματος αποκατάστασης προσφύγων. Θεωρούμε ότι αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό και θα συμφωνήσετε πιστεύω όλοι ε, σχετικά με το ότι ο φάκελος αυτός είναι κατεξοχήν φάκελος αλληλεγγύης ε, και ξαναλέω όχι μόνο ε, προς τα έξω αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. επαναλαμβάνω ότι πέρα από την πάγια συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, χρειάστηκε να επινοήσουμε ιδιαίτερα ε, φάνταστες ε, λύσεις για κάποια προβλήματα. Ελπίζω να συνεχίσουμε την αγαστή αυτή συνεργασία με τους δανούς φίλους μας. Ακολουθούμε πάντως κατά τη γνώμη μου το σωστό δρόμο. Κλείνοντας θα έλεγα ότι το... δεν είναι μόνο ενθαρρυντικό το ότι ακολουθούμε την σωστή ρότα αλλά ότι όλοι θεωρούν πως είναι κατεπήγον το ζήτημα. Αρχίζουν οι χώρες ε, να έχουν αξιώσεις για ε, ολένα και αυξανόμενο αριθμό προσφύγων τα κράτη-μέλη για να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τους νέου κανόνες όπω θα τροποποιηθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο του την επιπρόσθετα ε, κονδύλια ούτως ώστε να εντοπίσουμε ποια κράτη-μέλη δεν έχουν ε, παραδείγματο χάρη προγράμματα ε, αποκατάστασης προσφύγων ούτως ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να θεσπίζουν τέτοια προγράμματα για να αποκτήσουν αυτήν την συγκρηματοδότηση και για να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες ε, θα πρέπει να δράσουμε κατεπηγόντως. Ε, πιστεύω ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμμερίζονται αυτήν την άποψη ε, ήταν ομολογουμένως μακρόχρονη η διαδικασία είναι πάντως ε, πάρα πολύ σημαντικό που ξεκίνησε εγκαίρος, αλλά θα πρέπει να κλείσει και εγκαίρος ε, το θέμα της, ε, να ολοκληρωθεί η διαδικασία συναπόφασης. Ιδού. Α, ναι, σήμερα το απόγευμα προβλέπεται ο τριμερής διάλογος η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρέπει να κατοχυρώσει την εντολή ώστε να είμαι σε θέση να διαπραγματεύομαι με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επί τη βάση των ανησυχιών που ήγερα κατά τη διάρκεια τη παρέμβασή μα. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες, αλλά είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Θα έρθει και η κυρία Ρέντινγκ. Ε, την περιμένουμε στις 11, οπότε τώρα στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Σμιτ, και κατόπιν στον εκπρόσωπο του ε, Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεν ε, απέχουμε πολύ στην ουσία της πρότασης και δεδομένης και της σημασία του συγκεκριμένου ζητήματος, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, διότι όλοι όσοι συμμετέχουν θέλουν να ε, λειτουργήσει εγκαίρως αυτό το κοινό πρόγραμμα επανεκατάστασης, ώστε η διαδικασία του 2012 να υλοποιηθεί και βάσει των νέων κανόνων. Δράτω με της ευκαιρίας για να διορθώσω κάποιες πληροφορίες οι οποίες μόλις ακούστησαν. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Μαΐου, η διαδικασία δέσμευσης, επομένως έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε Εργαζόμαστε στενά ώστε να επιληθούν ε, όλα τα εναπομείνοντα προβλήματα και ελπίζουμε να υπάρξει επιτυχία στο τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, εκ μέρου του Συμβουλίου, η κυρία Κριστίνα Ρο από την Προεδρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο βλέπει θετικά τα τρία ζητήματα τα οποία έθιξε ο κύριο Ταβάρες στην ε, παρέμβασή του. Όσον αφορά την ανησυχία για το συνένα, δεν έχουμε άποψη επί του παρόντο για το θέμα αυτό. Πέραν αυτού, και εμεί ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το θέμα αυτό επειδή μα πιέζει και ο χρόνο και ανυπομονούμε να προχωρήσει ώστε να γίνουν οι δεσμεύσει πριν από την 1η Μαΐου ε, και τον καθορισμό των νέων κριτηρίων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να περάσουμε στο σκιώδη συγητή, τον κύριο Παπα-Νικολάου, εκ μέρους του ΕΛΚ. Just a short comment. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο. Ξεκινήσαμε τις εργασίες για το θέμα αυτό το 2010, είμαστε στο 2012, έχουν γίνει δύο-τρεις συζητήσεις ήδη, δεν θυμάμαι πότε, τρεις νομίζω στην Ολομέλεια, πολλές ε, προφορικές ερωτήσεις και προσπαθούμε συνεχώς να προχωρήσει το θέμα αυτό Το θέμα της επανεγκατάστασης ήταν ένα από τα πρώτα ζητήματα που είχαμε στην Επιτροπή μας εδώ στην Ολομέλεια μετά από την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Είχαμε κάποια προβλήματα διαδικαστικά και προσπαθήσαμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Η επανεγκατάσταση είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι κρίμα Και νομίζω αν δουν και οι πολίτες μας, οι ψηφοφόροι μας τι κάνουμε εδώ, δεν θα είναι και πολύ περήφανοι για μας διαπραγματεύομαστε για άλλη μια φορά ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό για ένα χρόνο μόνο, για το 2013. Μετά θα έχουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, νέες διαπραγματεύσεις ε, και ξανά μανά από την αρχή όλα. Ελπίζω να είναι τελευταία συνεδρία που θα κάνουμε για το θέμα αυτό. Α ελπίσουμε να το ολοκληρώσουμε και ο τριμερής διάλογος που θα γίνει το απόγευμα, α ελπίσουμε να είναι επιτυχής και να έχουμε καρποφόρα αποτελέσματα. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή, τον Ρουί Ταβάρες, για τις διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η μακρά διαδικασία. Ευχαριστώ εγώ κύριε Παπα-Νικολάου, η κυρία Νάντια Χίρς, σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Ρουί Ταβάρες για την εργασία του αλλά και για την αντοχή του όπως είπε και ο κύριος Παπα-Νικολάου προηγουμένως, ε, πολύ καιρό δουλεύουμε πάνω σε αυτό το ντοσιέ, σε αυτό το φάκελο, από το Φεβρουάριο. Μάλλον έχουμε φτάσει στο Φεβρουάριο και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε κάποια στιγμή. Και εμείς οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουμε απολύτως το Ρουί Ταβάρες ε, να διαπραγματευτεί τα θέματα αυτά. Ο κύριος Μπρόνσο. Ακούσαμε αναφορές από την Αίγυπτο, από την, ε, ε, την Ισία και από τη Λιβύη για τους ε, πρόσφυγες. Ε, ε, διέρχονται μια περίοδο εκδημοκρατισμού αυτές οι χώρες και οι πρόσφυγες όμως αυτοί κατέφτασαν στην Ευρώπη νωρίτερα κατά πάσα πιθανότητα. Ε, αν αυτό συμβαίνει, μήπως θέλουν να γυρίσουν και να προστατεύσουν τα νέα δημοκρατικά καθεστώτα αντί να είναι έγκλειστοι στους καταβλισμούς. Αν δεν ισχύει αυτό, από τι προσπαθούν να ξεφύγουν, από τη δημοκρατία. Εν τη αυτή περιπτώση θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους καλωσορίσει. Αναφερόμαστε επίσης σε πρόσφυγες από το Ιράκ και είπατε ότι δεν είναι όλοι Ιρακινοί, μπορεί να έρχονται και από αλλού δηλαδή. Ε, συγγνώμη, πού είναι αυτό το αλλού, ε, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν επικρατεί ασφάλεια στις άλλες χώρες από τις οποίες προέρχονται, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε κοινοτικά κονδύλια για να ε, επανεγκαταστάσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς τους πρόσφυγες και εφόσον μιλάμε για τους πρόσφυγες από το Ιράκ, θυμηθείτε ότι οι περισσότεροι από, αυτοί, από αυτούς τους πρόσφυγες ε, προέκυψαν από ένα ιδιαίτερα αιματηρό και καταστροφικό πόλεμο που ξεκίνησαν η ΙΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι. Ε, μήπως ε, ε, πριν ξεκινήσουν νέο πόλεμο κατά του Ιράν θα έπρεπε να τους θυμίσουμε τις ανθρώπινες επιπτώσεις, ε, τον αριθμό των θανάτων, τον αριθμό των προσφύγων που θα δημιουργήσει ένας νέος τέτοιος πόλεμος. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς, Χάνς και Αλφάνο. Σας παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα σύντομοι. Πάρα πολύ σύντομα υποστηρίζουμε και εμείς το Ρουίτα στο ε, στα μιλήματά του και στα τρία σημεία αυτά. Μπορώ να πω το εξή μόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι του Συμβουλίου, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε θετικά αυτό το θέμα. Καιρό είναι, σιγά σιγά αρχίζουμε και τρεπόμαστε που ασχολούμαστε τόσο καιρό με αυτό το θέμα. Thank no. Okay. Ευχαριστούμε κυρία Αλφάνο. Όχι, σβήνει το μικρόφωνο. Έχοντας ακούσει τον εισηγητή, του Σκιώδης και τους συναδέλφους, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια συνένωση για να δώσουμε προεντολή διαπραγματεύση ε, στον εισηγητή μας ε, για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Διαδικαστικώς πώς έχουμε περιορισμούς και είναι σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να καταρτήσουν τα σχέδιά τους για το 2013 βάσει της νέα απόφασης. Για να γίνει αυτό πρέπει ε, στη να ψηφιστεί ε, στην Ολομέλεια η απόφαση ε, το Μάρτιο σε περίπτωση θετικής έκβαση των συνομιλίων και διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο υπό το φω των σχολείων που έκανε σήμερα ο εισηγητή, αποσκοπούμε σε αποστολή επιστολή στην Κορεπέρε που θα αναφέρεται στο σημείο 18 της κοινή δήλωση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της διαδικασίας συναπόφασης για να ενημερώσουμε για ε, την ύπαρξη συμφωνίας. Δεν πιστεύω να έχει κανεί αντίρρηση για αυτή την επιστολή προς την Κορεπέρ. Πολύ ωραία. Ο εισηγητής θέλει να προσθέσει κάτι. Βλέπω μου ζητάτε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η κυρία Γκαμπρίλα Σμιτ ε, με διόρθωσε και καλά έκανα. Η διαδικασία pledging πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο η διαδικασία των αξιώσεων δηλαδή, και των δεσμεύσεων. Όταν ε, σας μιλάω για τη Λιβύη και την, ε, την Ισία, αναφερόμουν σε ε, ανθρώπους που προέρχονται από καταβλισμούς προσφύγων, που όμως συνήθως δεν έχουν την υπηκότητα της χώρας όπου βρίσκεται ο καταβλισμός. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαθιστά 4.500 ε, περίπου ε, πρόσφυγες και μιλάμε για τις πλέον, ξαναλέω, ευάλωτες ε, ομάδες προσφύγων. Και το ευχαριστώ. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος Επιτροπής μας θα αναλάβει και πάλι την Προεδρία. Yes. Thank you for your understanding. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Δεν μπορούσα να λείψω ε, τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας και Επίτροπε Ρέντινγκ. Έχετε το λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Ήγηκε η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό των όσων έχουμε επιτύχει και να δούμε και τι μας περιμένει. Όπως γνωρίζετε, το 2011 ήταν μια έντονη χρονιά. Σας κατέθεσα πάμπολε νομοθεσίες και έχουμε πάρα πολλές εντατικέ εργασίες εν εξελίξει ακόμα και ξέρω ότι η Επιτροπή σα ε, προσπαθεί να μας δώσει απτές ε, και καλές νέες πρωτοβουλίες για τις πολίτες μας. Να ξεκινήσω με τα πιο πρόσφατα τα οποία σας παρουσίασα την πρόταση μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Προστασίας Δεδομένων, την οποία ενέκνει η Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτούς της μεταρρύθμισης είναι να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα για την προστασία δεδομένων. Θέλουμε ο κόσμος να έχει έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων, ιδίως στο διαδικτυακό περιβάλλον, διότι όπως γνωρίζετε η παρούσα οδηγία είναι από το 1995, επομένως σε καιρούς προδιαδικτύου. Πώς μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να ανακτήσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να διευκρινίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κτήμα του καθενός. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος δίνει τα προσωπικά του στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώνεται για το τι ακριβώς θα κάνει μια επιχείρηση με τα δεδομένα αυτά και θα πρέπει να συμφωνήσει σε αυτούς τους κανόνες διαφάνειας. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να ανακαλέσει αυτά τα δεδομένα, την ε, ε, μεταφορά των δεδομένων. Το έχουμε κάνει και με τα ε, πακέτα των τηλεπικοινωνιών για τις δυνατότητες του τηλεφωνικού αριθμού. Όπως γίνεται λοιπόν ε, και με τις τηλεπικοινωνίες, μπορεί κάποιος να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων και να τα δώσει σε μια άλλη επιχείρηση. Ή μπορείτε και εσείς να τα ε, ανακτήσετε αν τα έχετε ξεχάσει. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή, αλλά αν συμβεί κάτι υπάρχει μια γενικότερη υποχρέωση να κοινοποιούνται παραβιάσεις δεδομένων είναι απαράδεκτο να χάνονται δεδομένα και οι καταναλωτές ε, να το μαθαίνουν τυχαία μερικές εβδομάδες αργότερα. Αυτά λοιπόν τα βασικά στοιχεία για τα προσωπικά δεδομένα. Θα εξορθολογήσουμε το ρυθμιστικό περιβάλλον. Μία Ήπειρος ένας κανόνας και μία ενιαία προσέγγιση για τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Ο επόπτης των δεδομένων θα είναι ο εθνικός επόπτης και θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους και ο εθνικός επόπτης θα αναλαμβάνει και τις ε, αναφορές και τις διαμαρτυρίες ε, του καθενός εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, ενός φυσικού προσώπου με μια επιχείρηση οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με υποστηρίξατε ιδιαίτερα στην ανακοίνωσή μου του 2011 για την προστασία δεδομένων. Υπήρχε και η σχετική έκθεση και είμαι πεπισμένη ότι και πάλι τώρα που έχει παρουσιαστεί ο κανονισμός θα ξεκινήσετε να εργάζεστε το στομότερο δυνατόν επ' αυτού. Στις 19 Μαρτίου θα υπάρξει μια διάσκεψη προστασίας δεδομένων στη Washington. Ε, από ό,τι κατάλαβα κάποιοι από εσά θα έρθουν στη Washington για να παρακολουθήσουν τη διάσκεψη αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί ε, το θέμα της προστασίας δεδομένων και με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και με τους εκπροσώπους που θα βρίσκονται στη διάσκεψη αυτή. Αναφέρθηκα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία ομπρέλα με την, για την προστασία δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενημέρωσα τους συντονιστές της Επιτροπής σας ε, για την κατάσταση αυτών των διαπραγματεύσεων αμέσως μετά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, νομένων Πολιτειών στο, στα τέλη του Νοεμβρίου του 2011. Στη συνεδρίασή μου με τους ε, ε Αμερικανούς ατέρους τους διευκρινίζω πάντα ότι το θέμα της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη δεν είναι υπόθεση, είναι προϋπόθεση, διότι είναι γεγραμμένο στις συνθήκες και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε όχι μόνο προς την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στην προστασία των δεδομένων εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Θα συνεχίσω λοιπόν να σας ενημερώνω συνεχώς επί της διαδικασίας και ε, θα σας ενημερώνω και αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη. Σε θέματα ποινική δικαιοσύνης. Η οδηγία για το δικαίωμα ενημέρωσης της ε, ποινική διαδικασίας εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και στην οδηγία για την ε, πρόσβαση σε ε, δικηγόρο, σε νομική συνδρομή. Διάβασα την έκθεση τη κυρία Αντωνέσκου και την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Άλμπρεχτ και νομίζω ότι λίγο πολύ ε, συνάδουν οι απόψει μας και ελπίζω να ολοκληρώσουμε σύντομα και ε, αυτό με πείθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δίκιο που πρότεινε υψηλά ποσοστά προστασίας για την προστασία των του καθενός και προσβλέπω και σε θετικά αποτελέσματα για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ακούσατε και τον Υπουργό Δικαιοσύνη της Δανίας, ήρθε και στην Επιτροπή σας και αναφέρθηκε και στο Ευρωπαϊκό Έντολμα Έρευνας, το οποίο θεωρεί προτεραιότητα για την Προεδρία του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει υψηλή ποιότητα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, να υπάρχει και αποτελεσματική έρευνα. Αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει επιτυχία επί του θέματος ε, και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθεια δική σας και της Δανικής Προεδρίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρω επίσης ότι σήμερα συζητήθηκε η έκθεση της κυρίας ε, Ρομέρο Λόπες, λέει ο Μιλήτρια, και της κυρίας Παρβανόβα για τα ε, ελάχιστα δικαιώματα θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Για το θέμα αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλα τα θέματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν βρίσκονται, έχουν κάποια ελάχιστα δικαιώματα και το βασικό δικαίωμα να τους συμπεριφέρονται ως ε, ανεξάρτητα άτομα και θα πρέπει να λαμβάνουν και την κατάλληλη ε, βοήθεια. Και για να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα για να, είναι πολύ σημαντικό για να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ενισχυθούν και τα μέσα προστασίας και τα μέτρα προστασίας και την αμοιβαία τους αναγνώριση. Και θα ήθελα να συγχαρώ τις κυρίες Παρμανόβα και Ρομέρο Λόπες για την έκθεσή τους. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά της έκθεσης θα μπορέσω να υποστηρίξω σίγουρα πολλά από αυτά και παρεπιπτόντως να σας ευχαριστήσω διότι αναφέρεστε και στις τοπικές αρχές οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, τα θύματα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Όσον αφορά τώρα τα ε, δικαιώματα ε, στη δίκαιη δίκη και δεν θα κάνω σχετικές προτάσεις επί του θέματος φέτος. Καταρχάς διότι θεωρώ ότι οι προτάσεις οι οποίες είναι ήδη επιτάπητος, ε, θα πρέπει να τεθούν πρώτα σε εφαρμογή και θα κάνω νέες προτάσεις το 2013, που είναι και το ευρωπαϊκό έτος ε, των πολιτών. Είναι το έτος ε, στο οποίο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επί τη βάση της πρότασης που τους έκανα πέρσι το θέμα αυτό και ξέρετε γιατί πρότεινα το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, διότι θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια δεν είναι κενό γράμμα, είναι μια ουσιαστική κατάσταση με ε, απτά αποτελέσματα ε, και σας ζητώ να εγκρίνετε τη σχετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το ευρωπαϊκό αυτό έτος. Δεν θα ήθελα να φτάσουμε στο 2013 και να ξεκινήσουμε τότε. Θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα το 2013 και να χρησιμοποιήσουμε και να υποφοληθούμε της εκστρατείας αυτής και για την ε, προεκλογική σας εκστρατεία το 2014. Θα ήθελα επίσης το 2012 να λάβουμε και τις ε, απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών για τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν ε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια εν γέννη. Θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε και την ατζέντα των πολιτών. Υπάρχει και η σχετική έκθεση για τους πολίτες ε, που θα, ε, θα παρουσιαστεί το 2013. Και επιτρέψτε με εδώ να σας πω και λίγα πράγματα ακόμα για τους πολίτες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τις πιο ευάλωτες ομάδες των πολιτών, όπως τους Ρωμά. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2011 έληξε με υπογραφή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπογραφή από όλες τις πλευρές, ότι θα προχωρήσουν και θα υπάρξουν εθνικές πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να ενσωματώσουν και αυτό το τμήμα του πληθυσμού στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Ήταν πολύ σημαντικό για την όλη διαδικασία. Υπήρξε και η έκθεση για Λούκα για την ενίσχυση της στρατηγικής ε, για την ένταξη των Ρωμά, η οποία αποτέλεσε έμπνευση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ε, ενσωμάτωση των Ρωμά, απασχόληση, ε, υγεία, στέγαση και παιδεία. Ξέρετε ότι αυτά είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία και τα συμπεράσματα τα επεσήμαναν αυτά τα στοιχεία. Πλέον εναπόκειται στα κράτη-μέλη για να καταρτήσουν την εθνική του στρατηγική. Μέχρι τούδε έχω λάβει 22 έγγραφα εθνικής πολιτικής Και αν ε, τα κράτη-μέλη δεν ε, εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, το γνωρίζετε ε, πάρα πολύ καλά ότι μπορώ να λάβω μέτρα. Τα πέντε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα προγράμματά τους έχουν κοινοποιήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα τα καταθέσουν εντός του Φεβρουαρίου, γεγονός που θα μου επιτρέψει από εκεί και πέρα τον Απρίλιο του 2012 να σας παρουσιάσω την έκθεση για τα 27 εθνικά προγράμματα δράσης. Προηγουμένως, στις 22 Μαρτίου, θα διοργανωθεί μια έκτακτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ένταξη των Ρωμά, ώστε να δοθεί δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να μας εκφράσουν την άποψή τους. Γνωρίζω ότι θα συμμετάσχουν αρκετοί από εσά ε, στην εκδήλωση αυτή. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η εκδήλωση. Ε, φαντάζομαι ότι θα είναι εκεί και η συγγήτρια και μου γνέφει καταφατικά, οπότε θα είναι παρούσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο πλαίσιο γνωρίζετε ε, πόσο σημαντική είναι η Οδηγία Ελεύθερης Μετακίνησης του 2004. Όταν θα εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία αυτή στα κράτη-μέλη, δηλαδή ο κάθε πολίτης, από όπου και αν προέρχεται, θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και φυσικά και θα έχει και τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά θα έχει τα δικαιώματα αυτά. Ξέρετε, του έδωσα μάχη με τη Γαλλία για το θέμα αυτό. Η Γαλλία αναθεώρησε την εθνική της νομοθεσία και έχει επιτεθεί σε ισχύ αλλά ενώ δινόταν η μάχη με τη Γαλλία, ανέλησε και πώ συμπεριφέρονται και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και διαπίστωσε ότι αρκετοί δεν έχουν εφαρμόσει καταλήλω την οδηγία του 2004. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε ένας διάλογος που σημαίνει ότι άρχισαν να πιέζω τα κράτη-μέλη ώστε να κάνουν αυτά τα οποία υποχρεούνται νομικώς να κάνουν. Και εάν δεν τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους, ξεκίνησαν διαδικασίες επί παραβάση. Οι περισσότεροι βέβαια ε, συμμορφώθηκαν, επομένως ε, έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, γίνει πραγματικότητα αυτό το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και με τις υποχρεώσεις και με τα δικαιώματα. Πάντα είναι δύο οι πλευρές του νομίσματος. Κατόπιν έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη αποτελούν υπόδειγμα σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τα θεσμικά του όργανα, οι θεσμοί τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό στην νομοθετική διαδικασία να εφαρμόζεται και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει το περιβόητο άρθρο 51 της Χάρτας που λέει ότι όπου ισχύει η Χάρτα ισχύει όταν νομοθετεί η Ευρώπη, αλλά και όταν εφαρμόζονται αυτοί οι ευρωπαϊκοί νόμοι από τα κράτη-μέλη. Ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόοδο σε αιτήσια βάση και ιδίω ο ρόλο που διαδραματίζει ο κάθε θεσμό, ώστε να φροντίσουν να συμπεριλαμβάνεται και αυτή η πτυχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε φορά που υπάρχει πρόταση για νέα νομοθεσία. Γνωρίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων για κάθε νομική απόφαση που λαμβάνεται. Δεν αφορά μόνο τους πολίτες και τις σχετικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και σε ε, οικονομικά, χρηματοπιστατικά ζητήματα ή οπουδήποτε αλλού. Η επόμενη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα εγκριθεί από την Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου. Αυτό για να ε, παραμείνει η όθηση που δημιουργήθηκε από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και προσβλέπω και στη συνεισφορά σας. Ξέρω ότι η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα θα α, αναλάβει το ζήτημα και θα το προωθήσει και εδώ. Τώρα, το πρόγραμμά μας. Στις 15 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο ε, προτάσεις ε, για να υπάρχει ένα πρόγραμμα δικαιοσύνης και ένα πρόγραμμα για τους πολίτες για το 2014-2020. Θα υπάρξουν ε, προτάσεις και χρηματοδότηση για την υλοποίηση των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Εξορθολογήσαμε και απλουστεύσαμε τα προγράμματα προκειμένου να υπάρχει προστιθέμενο όφελος Μέχρι τούδε υπάρχει πάγιος προπολογισμό για την ε, περίοδο 2014-2014, 911 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους δύο τομείς, με τρέχουσες τιμές. Είναι και πολλά και λίγα αυτά τα λεφτά, αλλά βασίζομαι σε εσά. Σε Ελπίζω να μην μειωθούν αυτά τα λίγα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε, όπως και στο παρελθόν, να υπάρχουν ομάδες υποστήριξης θυμάτων, ενημέρωση για το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπου υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετώπιση όλων των διακρίσεων ηλικίας, θρησκείας, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, καταγωγής, ε, οποιαδήποτε διάκριση λοιπόν υπάρχει, όλα αυτά σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με συνεχή τρόπο. Τέλος, η Ουγγαρία, γιατί ξέρω ότι θα γίνει και σχετική ακρόαση σήμερα το απόγευμα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, διότι θα σας δοθεί η δυνατότητα να τα συζητήσετε τα θέματα αυτά στη διάρκεια της ακρόασης, αλλά γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο και εγώ ενημερώσαμε την Ολομέλεια ότι έχουμε αποστείλει τρεις επίσημες επιστολές κοινοποίησης για θέματα δικαιοσύνης. Μία επιστολή σε θέματα αρμοδιότητας στο Ολιρέν για την Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας. Εγώ απέστειλα και μία εκ των προτέρων επιστολή για το άρθρο 258, ρωτώντας πληροφορίες για τη δικαστική δικαιοσύνη, ε, την ε, ε, λήξη της θητείας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίας, ε, τις εξουσίες του Προέδρου του Νέου Εθνικού Γραφείου Δικαιοσύνης και ούτω καθεξής, διάφορα τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, επομένως εντός ενός μηνός, δηλαδή στις 17 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν ληφθεί απαντήσεις. λαμβάνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις ε, οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένη νομική ανάλυση και ελπίζω ότι η Ουγγρική κυβέρνηση θα απαντήσει και θα μας προσκομίσει ε, τα στοιχεία και θα μας παρουσιάσει και τις ε, μεταρρυθμίσεις που σκοπεύει να κάνει. Ο πρόεδρος Μπαρόζο το διευκρίνησε αυτό και στον Πρωθυπουργό Ορμπάν στις 24 Ιανουαρίου. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι αυτά τα οποία ήθελα να πω εν είδη εισαγωγή. Σα ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ, για την παρουσίαση του προγράμματο εργασία στον τομέα τη δικαιοσύνη ε, για το επόμενο έτο. Ποια μέλη τη Επιτροπή θέλουν το λόγο. Κάνουμε το συνήθι πρώτο γύρο των συντονιστών καταρχάς. Να σας ενημερώσω όμως ότι μόλις με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα κρατικό πολωνικό, πολωνικό κανάλι που θέλει να κινηματογραφήσει ένα κλιπάκι από την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ε, έχει κάποιος ένσταση? Αλλιώς να τους δώσουμε την έγκριση για λίγα λεπτά να εισέλθουν στην αίθουσα και να κινηματογραφήσουν ε, ένα τμήμα της συνεδρίασής μας. Εντάξει, συμφωνείτε. Σάιμον Μπουζουτήλ. Φτιάξε και τη γραφάτα σου για την τηλεόραση. Um, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σας, για το έργο σας και για την υλοποίηση του προγράμματος στη Στοκχόλμη στην οποία προβαίνεται πρόγραμμα που είχαμε συμφωνήσει. Από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι της Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα σε σχέση με αυτό να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας υποστηρίζει και εσάς ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα κάνετε για την Ουγγαρία. Γνωρίζουμε ότι το κόμμα που κυβερνάει είναι κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αυτό μας κάνει να επιθυμούμε ακόμα περισσότερο ε, να τηρεί η χώρα τους κανόνες. Ε, διαδικασία προσφυγής ε, για τρία θέματα έχετε ξεκινήσει και ο δις από τον Πρωθυπουργό της χώρας ε, δήλωσε δημοσίω και στο Κοινοβούλιο μας ότι οτιδήποτε πρέπει να κάνει η ε, Ουγγαρία θα το πράξει, ε, ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς το κοινοτικό δίκαιο. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις και οποιασδήποτε αλλαγές πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στην νομοθεσία έτσι ώστε να συμμορφούνται πλήρως προς το κοινοτικό δίκαιο. Είναι λοιπόν αμέριστη υποστήριξή μας στο έργο σας. Ελπίζω όμως η συζήτηση αυτή να διατηρηθεί στο σωστό πλαίσιο, ε, ισορροπημένο και συγκρατημένο. Αν μια χώρα παραβιάζει τα καθήκοντά της με βάση το κοινοτικό δίκαιο, υπάρχει διαδικασία προσφυγής επί παραβάση ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία παρά να ε, κάνουμε απόπειρες να δημιουργούμε λαϊκά δικαστήρια που δεν μας οδηγούν πουθενά παρά μόνο στην πολιτική ε, αντιπαράθεση και στα παζάρια βασικά. Άλλα θέματα τώρα. Τα υπόλοιπα που αναφέρατε. Θα ήθελα να θυμίσω, μου επιτρέπετε, όπως έκανα και χτες, στη εφημερίδα Wall Street Journal. Χτες συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την εκπλήρωση της συνθήκης του Μαστρίχτ που όχι απλώς ελάνσαρε το εγχείρημα του ευρώ, αλλά και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. That I would like. Για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω και να επικεντρωθώ σε αυτή τη σχόλιά μου. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν αυτά Έγιναν πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αλλά ο κόσμο δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τι δικαιώματα έχει ω πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανεί και ίσω θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτά τα δικαιώματα και με νέα. Σα ερωτώ λοιπόν, το δικό σας όραμα ποιο είναι, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια για τους πολίτες μας τα επόμενα χρόνια, λαμβανωμένο υπόψη ότι του χρόνου θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Θαγένειας, αλλά επίσης και ε, ότι σήμερα είναι πολλές οι απειλές στην προώθηση ε, αυτής της ηθαγένειας. Κοιτάξτε τι γίνεται στη συζήτηση για το Σέγγεν, για παράδειγμα, που συνεχίζεται. Αν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να τα εξηγήσουμε αυτά με τρόπο εύληπτο και εύκολο για τους πολίτες, είναι ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας που υφίσταται τώρα επιθέσει από το Συμβούλιο. Άλλο παράδειγμα, οι θεωρήσει διαβατηρίων. Υποτίθεται ότι έχουμε όλη μια κοινή πολιτική, αλλά πολλές ε, τρίτες χώρες ακόμα κάνουν διακρίσεις ει βάρος των πολιτών ορισμένων ε, ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. And Αυτό θα πρέπει να είναι ένα τμήμα των όσων περιμένουν κανονικά από μας και από το διαβατήριο, όχι απλώς να αναφέρει τη χώρα του στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, αλλά να είναι ουσιαστική ε, η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το γράφει και το διαβατήριο, εκτός από το χρώμα. Λοιπόν, τι προτίθεστε να κάνετε. Η κυρία Μπόσκορτ από το Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την εισαγωγή της. Δεν καταλαβαίνετε Ολλανδικά, μάλλον δεν καταλαβαίνετε Ολλανδικά, υποθέτω. Βάλτε τα ακουστικά σας. Ωραία. Ε, Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχω και πολλές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις ακριβώς γιατί ασχολείστε με πολλά σημαντικά ζητήματα και ένα εξ αυτών είναι η τόσο απαραίτητη αναθεώρηση οδηγίας για την προστασία των δεδομένων με πολύ μεγάλη προσοχή θα το παρακολουθήσουμε, είναι απολύτως απαραίτητο. Έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση που αφορά αυτή τη δέσμη, ε, αλλιώς πακέτο των δικαιωμάτων των θυμάτων. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό στο Κοινοβούλιο ε, να ε, συμπληρωθεί και η διάσταση του φίλου Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το 2013 προτίθεστε να καταθέσετε νέες προτάσεις. Θα κάνετε ε, και πρόταση για θέματα φίλου. στη συνέχεια τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Πολύ σωστά σημειώσατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και να εφαρμόζεται. Συμφωνώ απολύτως. Αν κοιτάξετε την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί σας, τότε μας είχατε πει ότι, κοιτάξτε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Όταν ε, έχουμε ε, παντρεμένους ομοφιλόφιλους από την Ολλανδία, το Βέλγιο, άλλες χώρες που αναγνωρίζουν το γάμο, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αλλά δεν το εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη αυτό. Στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων έχετε υπόψη σα να κάνετε περαιτέρω βήματα το επόμενο διάστημα για να βελτιωθεί αυτή. Γιατί υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα και θα πρέπει να επιβάλλονται και να εφαρμόζονται και να έχουν τα ίδια δικαιώματα οι ομοφιλόφιλοι με τους ετεροφιλόφιλους. Άλλη ερώτηση. Τους transsexual. Πέρσι το κοινοβούλιο ζήτησε το Κοινοβούλιο να αφαιρεθεί ε, η περίπτωση αυτών των ατόμων από το χάρτη, από τον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών ε, για τις ψυχικές ασθένειες. οι transgender, οι διεμφυλικοί. Ε, γιατί έχουν πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού. Έχετε κάνει τίποτα, έχετε σκεφτεί καμιά πρωτοβουλία να το θέσετε υπόψη ε, στον ΠΟΕ, μάλλον στον ΠΟΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να αφαιρεθεί αυτή η περίπτωση από τα ψυχικά νοσήματα. Dat gaat over ε, de Άλλη ερώτηση. Οριζόντια οδηγία κατά ε, των διακρίσεων. Μας είπατε ότι στα νέα προγράμματα που ε, παρουσιάσατε στις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταπολεμείτε ε, η διάκριση ιδιαίτερα βάσει την ηλικία. Όλα αυτά είναι θαυμάσια, ωραία και καλά, αλλά έχει μπει στο ψυγείο αυτή η οδηγία. Μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm, is... Άλλο θέμα. Εκροδεξιά. Είχαμε το περασμένο διάστημα ε, πολλά παραδείγματα και πολλές ε, μελέτες που στοιχειοθετούν ε, ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά σε κάποιες χώρες όπως είναι η Γερμανία όπου έγινε η έρευνα, αλλά υπάρχουν ε, υποψίες ότι αυτό συμβαίνει και αλλού στην Ουγγαρία και τα λοιπά. Και επειδή η ακροδεξιά ε, απειλεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και κάνει διακρίσεις, έχετε κάνει τίποτα έρευνες για τέτοιου είδους τάσεις σήμερα στην Ευρώπη. Αυτά τα λίγα ερωτήματα και θα σας παρακαλούσα να μου τα απαντήσετε. Ευχαριστώ. Yes, please. Thank you. very much, Chairman, and thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο, διότι έκανε μια πληρέστατη επισκόπηση της κατάστασης ε, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ζούμε διαφόρων ειδών κρίσης. Η οικονομική κρίση μας οδήγησε σε κοινωνική και πολιτική κρίση και είναι πολύ πιο τρομακτικό το να διαπιστώνει κανείς όταν ταξιδεύει σε άλλα κράτη-μέλη ότι υπάρχει μια σχεδόν χαμένη γενιά νέοι ανεργοί που δεν έχουν απολύτως καμία ελπίδα ούτε και εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα ούτε και στους ερετούς εκπροσώπους. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ηθαγένεια. Η έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης ε, είναι κάτι που με τρομάζει πολύ περισσότερο από τις ε, διάφορες κρίσεις ε, που βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη. Τινούμε να ξεχνούμε δε ότι δεν είναι αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατά κύριο λόγο μια ένωση αξιών. Η αξιοπιστία μας η ίδια διακυβεύεται λοιπόν και αναφερθήκατε και το εκτίμησα στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως ε, η Ρωμά. Σας θαυμάζουμε, θαυμάζουμε το γνήσιο θυμό σας ε, όταν παρατηρήσατε ότι έγιναν αυτές οι μαζικές απελάσεις ε, από τη Γαλλία. Ε, όμως ε, περάσαμε κρίσιμους μήνες και είδαμε ένα, μια άλλη πολύ ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, αυτή τη φορά στην Ουγγαρία για να επανέλθω σε αυτή την κακόμερη χώρα. Το Δεκέμβρη πέρσι πέρασε ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου οι άστεγοι, οι φτωχοί, δηλαδή απροστάτευτοι και ευάλωτοι, ε, ποινικοποιούνται, ουσιαστικά ποινικοποιείται η φτώχεια τους. Ε, είναι εξαιρετικά ε, κοινικό και ιδιαίτερα τρομακτικό όταν αναλογιστεί κανείς ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ε, να ακούσω ποιο είναι το μήνυμά σας ε, χωρίς εξοραϊσμούς ε, σε σχέση με αυτό το φαινόμενο. Στην Ουγγαρία επλήγει λοιπόν αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Χτες δε έγινε ένα σεμινάριο για τους άστεγους στην Ευρώπη και σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν καθόλου στατιστικά στοιχεία για τους άστεγους. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, από 3 ως 5 εκατομμύρια στην Ευρώπη, είναι Ευρωπαίοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν λοιπόν ε, δεν θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον να χαρτογραφήσει την κατάσταση, να συλλέξει στοιχεία και να προτείνει έναν τρόπο ρύθμιση του προβλήματο, διότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, είναι συνυφασμένα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Οι φτωχοί που είναι άστεγοι σίγουρα δεν διαπράττουν κάποια αξιόπινη πράξη η έκτοτη ΕΝΔΕΗ στην Ουγγαρία σήμερα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο 455 ευρώ. Δεν θα έχουν αυτά τα λεφτά ή αλλιώς θα φυλακιστούν ή ε, θα κρατηθούν. Δεν ε, αντιδράσατε σε αυτό και θα ήθελα να κάνω ε, μία αντιπαράθεση με την κατάσταση των Ρωμά, γιατί είναι εξίσου σοβαρή η κατάσταση στην Ουγγαρία. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα ούτω ή άλλω το απόγευμα. Θα ήθελα όμω με σαφήνεια να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως τη δική σα άποψη, γιατί το έχετε ξανακάνει, σα εμπιστευόμαστε, έχετε ξαναπροστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα και αξίε στο παρελθόν με ε, τον πλέον κατάλληλο τρόπο ε, η ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα σε εσά και την Ουγγρική κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μα ε, δεν επαρκεί. Συμφωνείτε μαζί μου, Επίτροπε, ότι ένας επαγερός άνεμος φυσάει και διαπνεί την Ευρώπη και δεν σας μιλώ για την χαμηλή θερμοκρασία που είναι όντως ε, σχεδόν ανευπροηγουμένου, αλλά αυτό το ψύχος με τον, ε, σε συνδυασμό με τον ε, παγερό άνεμο μας έχει οδηγήσει σε καταστροφές. Επάνω από 400 άτομα πάγωσαν και πέθαναν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να επανορθώσετε την κατάσταση. Επανέρχομαι και πάλι στην Ουγγαρία που θα μας απασχολήσει το απόγευμα, ίσως όχι την παρουσία σας, Γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιες χώρες δεν θα επιτραπεί να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες τουλάχιστον. Αλλά όταν εισέλθει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται με αυτές τις ε, κυρώσεις για τι δίθεν αξιόπινες πράξεις. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτό. Θέλω μια αυθόρμητη αντίδραση. Δηλαδή ε, τίθεται να αμφιβόλο η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτε σε εμά. Και δεν σα μιλάω μόνο για τη χώρα μου, τη Σουηδία. Πήγα σε πέντε διαφορετικέ χώρες ε, τι προάλλε ε, στην Ευρώπη και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει φοβερή έλλειψη εμπιστοσύνη. Πρέπει να αιτιολογήσουμε τη συμπεριφορά μα και να ανταποκριθούμε στι ανάγκε των πολιτών, να επανορθώσουμε την κατάσταση, να διορθώσουμε ε, αυτά που κάνουμε και κυρίως αυτά που δεν κάνουμε. Ε, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερως αν μου δίνατε μια ειλικρινή απάντηση. Ευχαριστούμε κυρία Βίκστρομ. And, uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Αντιπρόεδρο για την ενημέρωση. <coughs> Υπόθηκαν ήδη πολλά. Θα επικεντρωθώ σε, of course, um, σε τρία πράγματα. Αναθεώρηση της ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Του καλωσορίζω. Πολλά από τα όσα αναφέραμε στην έκθεσή μας στην Περσινή έχουν υλοποιηθεί ήδη. Και ελπίζω πολύ σύντομα να αρχίσει η συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι. Γιατί πρέπει βεβαίως να διευρύνουμε τη συζήτηση ε, να δούμε τι προτείνει ο κανονισμός και η οδηγία για την αναθεώρηση τη προστασία των δεδομένων. Πάντως έχει νόημα, πιστεύω, πάρα πολύ σύντομα να αρχίσει η στενή διαβούλευση Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για να υλοποιηθούν, ε, να πραγματοποιηθούν αυτά τα δικαιώματα και να γίνει μεταρρύθμιση. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω, έχω και ερώτηση εδώ, είναι δικαστική συνεργασία. Είπατε ότι γίνεται συζήτηση για τα ελάχιστα ε, πρότυπα στην ποινική δικονομία. Έχουμε έκθεση της κυρίας Αντωνέσκο και το συζητούμε στην Επιτροπή μας. Συνεργαζόμαστε στενά για να διαμορφώσουμε κοινή θέση με την Νομική Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και ελπίζω αυτό να ε, γίνει προσεχώς. Um, Ερώτηση. Για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, ε, πραγματικά το συζητούμε και συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο γι' αυτό, αλλά τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από εκεί και πέρα είναι αντικείμενο συζήτησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, γιατί από πλευρά ε, Κοινοβουλίου ζητήσαμε λίγο να προσαρμοστεί σε σχέση με τη σημερινή του μορφή και θα παρακαλούσαμε να δραστηριοποιηθούμε σχετικά γρήγορα. Και ένα τελευταίο. η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Χάρτα, ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν γίνεται λόγος για ελάχιστα πρότυπα, θα πρέπει κάπου αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα να ε, μπορούν να εφαρμόζονται και να μπορεί κάποιος να προσφεύγει σε μια δικαιοδοσία για να γίνεται καλύτερη η διαχείρισή τους και να είναι καλύτερη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πολύ σημαντικό αυτό για μας όταν συντάσσουμε τέτοιες οδηγίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ελάχιστα πρότυπα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Επίτροπο διότι έκανα μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα και σφαιρική δέσμη προτάσεων αντιδρώντας σε πρόσφατες εξελίξεις. Ε, θα ήθελα να εστιάσω τις ε, παρατηρήσεις μου στον τομέα της συνεργασίας και πιο συγκεκριμένα στις ανησυχίες που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη λειτουργία των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Δεν αναφέρομαι στην Ουγγαρία εδώ, κάνω μια ευρύτερη αναφορά σε τομείς που ε, δεν ε, περιορίζονται σε κάποια οικονομικά συμφέροντα. Το λέω αυτό διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη της κυβερνοεγκληματικότητας ε, και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη δράση σε αυτό το τομέα. Είναι βασικό θέμα ακόμη και όταν κάποιος όπως εγώ ε, σέβεται τα εθνικά ποινικά συστήματα των κρατών μελών όπως κάνει φαντάζομαι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Παρόλα αυτά, σε κάποιους τομείς πιστεύω ότι είναι απόλυτα ορθό και θεμητό να περιμένουμε από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίζουν πρότυπα τα οποία τουλάχιστον συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο ή ε, τις διεθνείς συμβάσεις. Το θέμα των όρων υποδοχής των ετούντων άσυλο είναι ένα ζήτημα που με έχει αποσχολήσει επανειλημμένα και στο παρελθόν και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω μια βαθιά ανησυχία την τελευταία φορά που προσπαθήσαμε να αναδιαπραγματευτούμε για το Δουβλίνο, τον κανονισμό Δουβλίνο, και συνειδητοποιήσαμε ότι πραγματευόμαστε με, πρέπει να πραγματευόμαστε μάλλον με ορθό τρόπο τις αιτήσει ε, ασύλου Διαπιστώσαμε ότι σε διεθνέ επίπεδο τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούνται ω ασφαλεί χώρε όπου ε, κάποιο ευχερό μπορεί να αιτηθεί άσυλο. Όπως σας έλεγα, ε, δεν επιθυμώ να παρεσφρείω σε εθνικά συστήματα ποινικού δικαίου, αλλά εδώ διαφέρει η κατάσταση και δεν θα ήθελα να επαναληφθούν καταστάσεις, επίτροπε, όπως ε, άνθρωποι που είναι στη Γερμανία, στη Βρετανία ή αλλού, δεν έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν, να επαναπροωθηθούν σε άλλες χώρες λόγω των προτύπων που ισχύουν στην Ένωση. Ρωτώ το εξή. Όταν εξετάσετε εξετάζετε το θέμα των δικαστικών ζητημάτων και της ε, Δικαστική συνεργασία ε, και αυτή η συνεργασία ε, δεν είναι μονόδρομος, ε, πρέπει να είναι αμφίδρομη η συνεργασία και με την διεθνή κοινότητα ως προς τα πρότυπα που εφαρμόζουμε στον τομέα αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να προσθέσετε, Επίτροπε, κάτι παραπάνω για αυτό το ζήτημα πριν αποχωρήσετε. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Έρνστ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντιν, καταρχάς για την παρουσίασή σας, για τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Και νομίζω ότι όντως είναι το σωστό πρόγραμμα για το 2012. Αυτό που μας παρουσιάσατε για την αρμοδιότητά σας και σας υποστηρίζουμε πάρα πολύ στεναρά. Έρχομαι τώρα σε μερικά θέματα που με απασχολούν και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και πάλι η Ουγγαρία. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ επίμαχη και συγκρουσιακή και θα συνεχιστεί και το απόγευμα, ούτε πρόκειται να σταματήσει πιστεύω. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και εσεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κοιτάξουμε τι γίνεται με το κοινοτικό δίκαιο και πόσο το δίκαιο της χώρας ε, συμμορφώνεται προ αυτό. Αλλά γνωρίζουμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο, ότι είναι βαριά παραβίαση του κράτου δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω πάρει πολλά μηνύματα από οργανώσεις και γράμματα ε, οργανώσεις ομοφιλοφίλων στην Ουγγαρία που ανησυχούν πάρα πολύ και λόγω ε, του νέου οικογενειακού δικαίου που εγκρίθηκε τώρα στην ε, Ουγγαρία και έχουν, ας πούμε, ο Κρίστοφερ Στρίτ έχει πρόβλημα να βγει στο δρόμο. Γιατί οι, ε, αστυνομικοί που υποτίθεται ότι τους φρουρούν, ότι τους φυλάτουν, μπορεί να είναι ακροδεξιοί και να τους απειλούν. Αυτό το λένε πολλοί. Ε, ε, Ουγγροί ομοφιλόφιλοι δεν τολμούν να βγουν να διαφυλώσουν το δρόμο. Τι θα κάνετε για να προχωρήσουμε εκεί σε αυτό το θέμα και την καταπολέμηση της διάκρισης των ομοφιλοφίλων. Ε, Προστασία δεδομένων και μεταρρύθμιση αυτής. Χαίρομαι πολύ που ε, υιοθετήσατε τις προτάσεις μας που εμείς καλωσορίζαμε και προωθούσαμε και είναι πολύ ε, θετικά όλα αυτά που μας προτείνετε. Στη Γερμανία γίνεται μια συζήτηση. Τι γίνεται με τις ρυθμίσεις ε, που είναι υπερκείμενες των ελαχίστων προτύπων. Ας πούμε ότι έχουμε θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν αυστηρότερη νομοθεσία. Στη Γερμανία γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και εγώ διαρωτώ με και σας ρωτώ και σας ε, ευθέω, γιατί δεν έχετε από την αρχή ε, διευρύνει ε, τις ε, προτάσεις σας για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι πολλοί κόσμος, χιλιάδες. Γιατί το έχετε εξαιρέσει αυτό το σχέλος Ρωμά, τι άλλο. Άλλωστε, πέρσι το Δεκέμβριο στο Βερολίνο είχαμε ένα συνέδριο που συμμετείχαν Ρωμά από 15 χώρες και συνεχώς ε, μας μιλούσαν για τη στρατηγική που εγκρίναμε ε, ότι η στρατηγική μας πραγματικά ε, προχωρεί με βήμα σημειωτών. Δεν κάνει μεγάλα βήματα και λένε επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχετε τις εθνικές στρατηγικές, τις αναλύετε και αν έχουν αποτελματωθεί, τι σχεδιάζετε, κατά τη γνώμη σας τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά τα θέματα. Και ένα τελευταίο πρόβλημα. Εγώ προέρχομαι από εκείνο το κρατήριο της Γερμανίας που ε, έδρασε ε, η περίφημη αυτή ναζιστική ομάδα και ε, σκότωσε, δολοφόνησε πολίτες στη Γερμανία. Είναι νεοναζί αυτή και με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του νεοφασισμού και της ακροδεξιάς. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει εδώ να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία, ενδεχομένως και με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που θα πρέπει να ενέχεται πολύ πιο έντονα, για να αποτρέψουμε την προέλαση της ακροδεξιάς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά στην Ευρώπη. Now, I have not noticed any further hands, particularly for the δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Για τον πρώτο γύρο των συντονιστών ε, δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο πλευράς της ομάδας EF2, οπότε... Ε, θέλουμε ούτως ή άλλως να ακούσουμε τις απαντήσεις της κυρίας Ρέτινγκ στις ερωτήσεις των συντονιστών και μετά θα κάνουμε δεύτερο γύρο για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ε, ε μάλλον τους υπόλοιπους βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Ρέντινγκ. Θέλω να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, τα, τους βουλευτές, διότι έθεσαν πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα και πολύ άριθμα, κυρίως για την Ουγγαρία. Ε, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, μπορεί να παρέμβει μόνο σε θέματα νομοθεσία της Ένωσης. Η Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Δεν μπορεί να υπερβεί ε, την συνθήκη, λειτουργεί μόνο μέσα στα όρια της συνθήκης. Πέρυσι, ε, διάφορα προγράμματα δρομολογήθηκαν και εγώ ε, συνέταξα μία επιστολή την ανέφερε και η, η Υπουργός Κλίντον στη δική της επιστολή για αυτό το θέμα της Ουγγαρίας υπάρχουν ε, ε, ε, τίθεται ζήτημα συνταγματικής τροποποίησης και αν τα προτινόμενα νομοσχέδια ευθυγραμμίζονται ή όχι με την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης. Αυτό ήταν το ζήτημα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση εξάλλου μπορούμε να παρέμβουμε. Αν αντιβαίνουν αυτοί οι νέοι νόμοι στην νομοθεσία της Ένωσης. Δεν μπορούμε όμως να επέμβουμε όταν μια νέα νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο δεν βασίζεται, δεν εδράζεται, αν θέλετε, στο, δευτερογενές, στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο της Ένωσης. Σε Κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν αυτό, διότι θα μπορούσαμε ε, να επέμβουμε ενδεχομένω και σε υποψήφια για προσχώρηση χώρα. Όμως δεν μπορούμε να παρέμβουμε όταν μια χώρα έχει γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να κάνουμε έτσι προβλέπει ο νόμος. Ο Σάιμον Μπουσουτήλ παρέθεσε απόσπασμα από το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Wall Street Journal και προτείνω σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο οδικό χάρτη για θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί λοιπόν αυτός ο οδικός χάρτης. Είδαμε, διαπιστώσαμε ποιες είναι οι ατέλειες και νομίζω ότι όταν διαπιστώσουμε όλες ε, οι αδυναμίες, όλα τα κενά που ακριβώς βρίσκω, θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και μία διάσκεψη, ούτω ώστε να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο και να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως παραδείγματος χάρη και τώρα θα ε, ε, επανέλθω στο ερώτημα της κυρίας Μποσκούρτ, ε, για θέματα οικογενειακού δικαίου να ξέρετε ότι είναι αδύνατη η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά που, οι προτάσεις που κατέθεσα τώρα έχουν ως στόχο μεταξύ άλλων να υπερκεράσουν αυτές τις δυσκολίες, να γεφυρώσουν τα κράτη-μέλη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προσπαθώ να επέμβω σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Με ρωτήσατε αν αληθεύει ότι 20 χρόνια μετά την θέσπιση της έννοιας ε, της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συνθήκη του Μάστριχτ παρόλα αυτά δεν υπάρχουν δεν υπάρχει ενημέρωση και γνώση των δικαιωμάτων της, ε, ε, που επισύρει η Ιθαγένεια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν θα είναι τόσο σημαντικό το 2013 που θα είναι έτος Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Για διάφορους λόγους πρώτον θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που επισύρει η Ιθαγένεια και στη συνέχεια θα ρωτήσουμε τους πολίτες τι πιστεύουν σε σχέση με την καθημερινή εφαρμογή, ε, άσκηση μάλλον των δικαιωμάτων τους ε, στα κράτη-μέλη. Θα δράξουμε την ευκαιρία αυτού του ευρωπαϊκού έτους και ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο. Έχω επίσης εισηγηθεί Παραδείγματο χάρη, σε αυτό το πλαίσιο, ε, τα νέα δικαιώματα ως προς την προξενική προστασία. Και θα με ικανοποιούσε πολύ αν προωθούσατε κι εσείς αυτό το θέμα, διότι ε, θεσπίζονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, νέα δικαιώματα, ούτως ή άλλως ε, στην προηγούμενη συνθήκη ήδη είχε γραφεί η ιδέα, τώρα έχουμε περάσει την πρακτική εφαρμογή, έκανα και εγώ την εισήγησή μου, βοηθήστε με σας παρακαλώ, ούτως ώστε να μπει στις δράγεις και να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Ο κύριος Μπουζουτήλ μίλησε επίσης για απειλές στο χώρο του Σέγγεν, για τις θεωρήσεις, κυρίως για το Σέγγεν. Ναι, σας απαντώ ότι ανησυχώ, όπως και πολλοί από εσάς, για τον τρόπο με τον οποίο ε, ασαφείς κανόνες ή τουλάχιστον κανόνες που δεν είναι ε, εναργείς χρησιμοποιούνται για άλλους πολιτικούς ε, στόχους με πλημελή τρόπο. Υπάρχουν καταχρήσεις και αυτό το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Γι' αυτό και η συνάδελφος Σεσίλια Μάλμστρεμ εξεργάζεται προτάσεις ε, για να βοηθήσει αυτά τα που κάνει θα δώσουν την απάντηση, πιστεύω. Υπάρχουν βεβαίω, από ό,τι ξέρω, πολλά κράτη-μέλη που αντιτίθενται στη θέσπιση εναργέστερων κανόνων ω προ την κινητικότητα των πολιτών και όταν ετέθη το ζήτημα, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης, το χώρο του Σέγγεν, επενέβη ε, παραδιαφόρων ε, υπουργών για να διευκρινίσω ότι θα αναλάβουμε δράση ούτως ώστε ε, να μην κινδυνεύουν και να εφαρμόζονται σωστά στην πράξη και να ασκούνται σωστά στην πράξη τα δικαιώματα των πολιτών. Κύριε Μποσκούρ, θέσατε διάφορες ερωτήσεις για ζητήματα που άπτονται τις ισότητες των δικαιωμάτων των δύο φύλων. Η πρώτη σας ερώτηση σχετιζόταν ε, με τις ε, γυναίκες ε, και τη βία. Το πακέτο για τα θύματα είναι ουδέτρο από πλευράς φύλου. Όπως ακριβώς και οι δύο εντολές προστασίας. Αυτοί που θα υποφεληθούν περισσότερο σε εισαγωγικά, αυτοί δηλαδή που θα επικουρηθούν από το ένταλμα, ξέρετε, θα είναι κατεξοχήν οι γυναίκες και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ένα άλλο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας. Η κυρία Χιμένες Εμπεσερίλε και η κυρία Παρβάνοβα προσπαθούν να οριοθετήσουν ε, ε, τις ευάλωτες, ε, τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες θυμάτων. Θα δείξω ανοιχτό πνεύμα και θα συζητήσω τις νέες προτάσεις τους μαζί τους για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων θα ήθελα να πω το εξής. Ε, ε, να γνωρίζετε ότι ολόκληρο το ζήτημα της ισότητας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, όχι μόνο λόγω φύλου, λόγω ηλικίας και ούτω καθεξής, είναι ένα θέμα που εντάσσεται και στην οδηγία για την κατάργηση της ε, διακριτικής μεταχείρισης, όμως μόνο στο χώρο εργασίας. Η διακριτική μεταχείριση εκτός ε, εργασιακού χώρου έχει παγώσει ε, στο Συμβούλιο. Κάθε φορά που πάω στις χώρες που παγώνουν τη διαδικασία και συναντιέμαι με τους υπουργούς τους, επαναφέρω στο τραπέζι το θέμα. Δυστυχώς δεν κατάφερα να απεμπλέξω την κατάσταση. Η περίφημη οδηγία του άρθρου 19 δεν υπάρχει πουθενά λοιπόν. Τι έκανα στο ενδιάμεσο διάστημα παρόλα αυτά. Ακριβώς διότι δεν μπορώ να επέμβω σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου στα κράτη-μέλη αν παρεμβαίνω αλλού και πού μπορώ να παρέμβω σε ζητήματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κατέθεσα διάφορα σχέδια νομοθετημάτων, παραδείγματος χάρη για τους διεθνείς γάμους και διεθνή διαζύγια ή ε, για την κληρονομική διαδοχή ή για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των εγγράφων. Όλα αυτά είναι ουδέτερα από πλευράς φύλου. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα που θεσπίστηκαν σε ένα κράτος μέλος, όταν οι άνθρωποι επί τη βάση αυτών των δικαιωμάτων εκμεταλλεύονται την ελευθερία μετακίνησης ε, πρέπει να γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα από όλες τις χώρες τις οποίες ε, ε, ταξιδεύουν. Είμαι σίγουρη ότι θα με βοηθήσετε να συνεχίσω τη δουλειά για όλα αυτά τα σχέδια νομοθετημάτων, διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και εξάλλου εκεί έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, όλο αυτό το θέμα των ε, εξτρεμιστικών κινημάτων ή οργανώσεων. Είδαμε όχι μόνο στην Ουγγαρία, στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ε, τέτοια κινήματα. Διαπιστώσαμε την ύπαρξή τους και σε άλλες χώρες και ενισχύονται διαρκώς ε, λόγω της ε, μεγέθυνσης των οικονομικών προβλημάτων. Οι άνθρωποι φοβούνται και υιοθετούν ακραίες ε, θέσεις ακριβώς λόγω του φόβου αυτού. Και πάλι εδώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου και βοηθά τις ε, κυβερνήσεις που επί τη βάση του συντάγματος τους ε, συζητούν αυτή τη στιγμή αν ε, πρέπει να απαγορεύσουν ή όχι τέτοιου είδους κινήματα. Όταν βλέπω τις συζητήσεις που γίνονται στη Γερμανία παραδείγματος χάρη διαπιστώνω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να απαγορευτεί ένα κόμμα ή ένα κίνημα χρησιμοποιώντας ως νομική βάση το σύνταγμα της χώρας. Γίνονται σοβαρότατες συζητήσεις λοιπόν από αυτού και είναι σημαντικό να τροφοδοτήσουμε και εμείς αυτές τις συζητήσεις και να αναδείξουμε όσο ε, σημαντικό και το θέμα των δικαιωμάτων. Αυτό με φέρνει και στην ερώτηση της κυρίας ε, Βίκστρομ για την χαμένη γενιά, την κρίση, το, τα εξτερμιστικά κινήματα, την απώλεια εμπιστοσύνη και αξιοπιστίας. Κυρία Βίκστρομ, απολύτως δίκιο έχετε, όπως και άλλοι συναδελφοί σας. Όταν ε, δείτε τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου θα διαπιστώσετε ότι με τα χρόνια καταμετρήσαμε αναέτος ε, την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες ε, στα, στις χώρες τους, στις κυβερνήσεις τους και στη, στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Κατά μέσο όρο ε, ήταν μάλλον σταθερή αυτή η εμπιστοσύνη και είναι λίγο υψηλότερη η εμπιστοσύνη που έχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτή που έχουν στι εθνικές κυβερνήσεις. Κατά μέσο όρο το τονίζω και δεν ισχύει αυτό για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά είναι ενδιαφέρον ε, σημείο εκκίνησης ε, και θα ήθελα να σας πω ότι ε, η εμπιστοσύνη τώρα αυθύνει. Ευθύνη και ευθύνη σε σχέση με τους πολιτικούς ηθήνοντες σε εθνικό επίπεδο. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η τάση και για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία στην Ευρώπη. η απόδειξη της εμπιστοσύνης μέσα από μια διαδικασία ψηφοφορίας, η εμπιστοσύνη ότι ε, κάποιος θα επιτελέσει κάποιες ευθύνες εξ ονόματος του λαού, αυτή είναι η βάση της δημοκρατίας. Αν αθετηθεί αυτή η υποχρέωση, τότε θα έχουμε τέτοιου είδους ε, προβλήματα και θα υπάρξουν προβλήματα στις διαδικασίες επιτέλεσης των καθηκόντων μας ε, κυρίως μιλώντας για τους ερετούς εκπρόσωπους του λαού και νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ε, ε, συζήτησης στο Κοινοβούλιο γιατί είναι θέμα δημοκρατίας ε, και ξέρετε όταν πηγαίνετε σε μια χώρα και συναντάτε ανθρώπους μπορεί να θεωρήσετε ότι όλα αυτά δεν είναι σημαντικά. Όταν βλέπετε όμως το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωβαρόμετρο, ε, διαπιστώνεται πόσο ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις. Οι ευάλωτοι συμπολίτε μας όπως η Ρώμα προστατεύονται, κάνουμε αρκετά ή όχι, θα μπορέσουμε κάποτε να κάνουμε αρκετά, διότι μόνο η δράση μας περιορίζεται από τις αρμοδιότητες που έχουμε και γι' αυτό θα επανέλθω στους τέσσερους πυλώνες. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει γραπτός και με σαφήνεια να καταθέσουν τα εθνικά σχέδια δράσης τους ούτως ε, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι. Δεν μπορούμε να ε, περιοριζόμαστε σε γενικόλογες ε, συζητήσεις και αυτό το λέω σε σχέση με την οδηγία που κατοχυρώνει ελεύθερη κυκλοφορία. Γιατί έτσι μπορεί να γίνουν προσφυγές κατά κρατών μελών. Όμως, Ε, η οδηγία δεν εξασφαλίζει ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία σε επίπεδο κράτους μέλους. Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια, ξέρετε, για να εφαρμόσουν ε, αυτούς τους κανόνες ε, και πάλι εδώ οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη ότι πολλοί δεν αγνοούν αυτά τα δικαιώματα, δεν ξέρουν καν ότι έχουν δικαιώματα. Γι' αυτό και είναι καλό το 2013 το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας για να δώσουμε διευκρινήσεις. Θα σας εξηγήσω δε στην Ολομέλεια ελπίζω ε, ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα και κάθε χρόνο θα διεξάγουμε ανάλυση των πεπραγμένων γιατί η κατάσταση των Ρωμά δεν επιλύεται, δεν ρυθμίζεται σε ένα δεκαπενθήμερο. Είναι μια μακροχρόνια επένδυση και γι' αυτό το λόγο πέμενα να πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, διότι πρέπει να λύσουμε ακριβώ αυτό το πρόβλημα των μελλοντικών χαμένων γενεών. Θα δούμε την ανάλυση της κατάστασης στα 27 κράτη-μέλη, θα υποβάλουμε την έκθεση και θα έρθω στην Ολομέλεια και να σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα. Το θέμα των αστέγων και η ποινικοποίηση της ένδυας. Είμαι ε, χριστιανοδημοκράτης, ε, και δεν έχω πρόβλημα με τέτοια θέματα, αλλά αυτές είναι οι προσωπικές μου απόψεις. Έχουμε εμεί ε, δικαιοδοσία αρμοδιότητα για ε, τέτοια νομοθετήματα. Θα πρέπει να συνομιλήσω με τον συνάδελφο αρμόδιο για τις κοινωνικές υποθέσεις για να διαπιστώσουμε αν ε, προβλέπεται αρμοδιότητα της Ένωσης στο τομέα, της Επιτροπής στον τομέα αυτό. Ε, ούτως ή άλλως, κάτι που ήδη κάνω με συστηματικό τρόπο και σε όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως ε, στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει πρόβλημα είναι το εξή. Ενίσχυση των δικαστηρίων, ούτω ώστε να επικρατήσει νομική ασφάλεια και οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν ενώπιον του δικαστηρίου όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, σε σχέση με την επιστολή που στείλαμε στην Ουγγρική κυβέρνηση, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ζητήσαμε πληροφορίες, διότι χρειαζόμαστε αμερόληπτο δικαστικό σύστημα και το δικαίωμα της αμερόληπτης διοίκησης εγγράφεται στη Χάρτα Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να εφαρμοστεί κιόλα, διότι ήδη υπάρχει στο συνολικό πακέτο των ε, δικαιωμάτων το απόγευμα στην ακρόαση που θα γίνει ο Γενικός Διευθυντής η Γενική Διευθύντρια μου μάλλον θα έρθει και θα είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, είναι σε θέση να με εκπροσωπήσει πλήρως. Δεν έγινε ανταλλαγή επιστολών με την ε, Ουγγρική ε, κυβέρνηση. δεν έκαναμε μια απλή ανταλλαγή επιστολών. Τι θες, προσφυγής. Ή τροποποιείτε την νομοθεσία σας ή θα ε, επιληφθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ε, εντολή ε, προστασίας. Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και όλα τα Όλες οι επιμέρους συνιστώσεις ε, πρέπει να συζητηθούν ε, διότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα γενικό που καλύπτει διάφορες διαστάσεις της πολιτικής. Ε, δικαστική συνεργασία και τώρα επανέρχομαι σε διάφορα ερωτήματά σας. Είναι εκ των ουκάνευ ε, να κατοχυρώνονται τα ελάχιστα δικαιώματα μέσω της δικαστικής συνεργασίας για όλους. Παρότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι πιο ισχυρά από αυτά τα δικαιώματα, μάλιστα. Αλλά τουλάχιστον τα ελάχιστα δικαιώματα είναι σημαντικά και για την εντολή έρευνας ε, και έλαβα το μήνυμα ότι θέλετε να συνεργαστείτε με τη Δανική Προεδρία για αυτό το θέμα. Τώρα, το ένταλμα σύλληψη. Κάναμε τη συζήτηση αυτή ήδη στην Ολομέλεια. Πολλά είναι τα προβλήματα. Όχι με το ένταλμα σύλληψη αυτό καθευτό, αλλά με την ε, εφαρμογή του. Διότι κάποια κράτη-μέλη κάνουν καταχρήσεις για μικροπαραβατικότητα, μικροεγκλήματα. Δεν είναι για παραπτώματα, είναι για ε, ε, ε, σοβαρές αξιόπινες πράξεις, κακουργήματα, όχι να κλέψει ένα κοτόπουλο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Έστειλε επιστολή σε όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης να το εφαρμόσουν σωστά, όχι για πτέσματα και να μην προχωρούν σε καταχρήσεις γιατί αυτό θα καταστρέψει την όλη προσπάθεια. Τώρα το θέμα της ε, προσχώρηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την ΕΣΔΑ. Εγώ έχω εντολή για να κάνω διαπραγματεύσεις. Τι ολοκλήρωσα. Πάρα πολύ δύσκολε, οφείλω να σα πω. Ε, θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα όπου το ΔΕΚ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου να αλληλοσυμπληρώνονται και να μην ε, αλληλοπλοκάρονται. Τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει να τα κυρώσουν όλα αυτά. Αυτό είναι το θεμα Τα Ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν να κυρώσουν τέτοιες ε, συμφωνίες και την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ. παρόλο που δεν είναι δυνητική αυτή η ε, διάταξη, είναι υποχρεωτική, την περιγράφουν οι συνθήκες. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως βλοκάρουν ε, διότι δεν θέλουν απλούστατα να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ε, Council of Ministers now is presided by Great Britain. Τώρα, ας πούμε, όπως αποφάσισε η Μεγάλη Βρετανία, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει, αν θα εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα που προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών και θα κάνει μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, στο δικαστήριο. Είναι πάρα πολλά τα αδιέξοδα. Θα ήταν σημαντικό, λοιπόν, να ε, προωθηθούν κάποιες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Ζητώ, λοιπόν, δημόσια από ε, τη Βρετανική Προεδρία που προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργό τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να φανεί χρήσιμη. Αυτό θα μα εξυπηρετούσε πάρα πολύ και θα ήταν ιδιαίτερο θετικό. Η ε, Διεθνή δικαστική συνεργασία, ε, κύριε Κίρκοπ, και οι εθνικέ διαφορέ βεβαίω είναι δεδομένε αυτέ. Και δεν μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε τα εθνικά συστήματα των χωρών. Κάθε χώρα έχει το σύστημά της και αυτό είναι ευθύνη της εκάστοτε χώρας, του εκάστοτε κράτος. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ για τα διασυνοριακά να έχουμε ελάχιστους κανόνες και να δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Τα κράτη-μέλη μας συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του διεθνούς δικαίου. Αξιότιμη κύριε Κύρκοπ. Τα εθνικά δικαστήρια μας έχουν δώσει σαφέστατη αρνητική απάντηση. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί η έκδοση προς ορισμένα κράτη-μέλη. Και την υπόψη στην Ελλάδα προφανώς, ναι. Έχουμε τους εμπειρογνώμονές μας, εμείς ποιοι είμαστε εμείς. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης έχει στείλει εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα για να βοηθήσει να μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα. Ε, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί στην Ελλάδα όσα όφιλε, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα και ε, όχι σε ασφάλεια δικαίου. Θέλουμε να βοηθήσουμε ε, ε, την Ελλάδα να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και για την αστική δικαιοσύνη και για άλλα θέματα, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη που χρειάζεται οπωσδήποτε ε, να επανέλθει σε όλα τα κράτη-μέλη. Γενικώ βεβαίως ανησυχούμε. για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία για το άσυλο και η σύμβαση του Δουβλίνου. Η συνάδελφο Σεσίλια Μάνστρομ ε, εργάζεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απογοητευμένη. Δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά της για να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να βοηθήσει και η Επιτροπή σας αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Ένστ ρώτησε για την Ουγγαρία. Το οικογενειακό δίκαιο, το απάντησα αυτό ήδη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές βάσει των ε, δικαιωμάτων που συμφωνήσαμε από κοινού. Κάθε φορά που είχαμε μεγάλες διακρίσεις, ας πούμε, απαγόρευση ε, των παρελάσεων, όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και αλλού, Προσπάθησα κάθε φορά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε ε, στις ευρωπαϊκές μας αξίες διακρίσεις. Προστασία των δεδομένων. Αυτό το είναι γερμανικό ζήτημα. Κοιτάξτε, ανέλησα τους κανόνες που ισχύουν για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα διάφορα κράτη-μέλη εμπνεύστηκα από τα καλύτερα κράτη-μέλη και υιοθέτησα τις βέλτιστες πρακτικές και ε, τις εισήγαγα σε ένα ευρωπαϊκό κανόνα και ε, όλα αυτά επεκτάθηκαν και στα άλλα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό. Η Γερμανία που έχει πολύ ισχυρούς κανόνες θα δει τους κανόνες αυτούς να καθίζονται ευρωπαϊκοί. Και αυτό είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε, ε, να αρχίσουμε από το υψηλότερο δυνατό κατόφλι. Και είμαι βεβαία ότι στις συζητήσεις που θα κάνει το Κοινοβούλιο στο μέλλον θα διατηρήσει αυτό το υψηλό κατόπιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όπως σας είπα και σήμερα το πρωί, έχουμε φρικτό πρόγραμμα για σήμερα. Έχουμε προγραμματίσει στις 12.30 να κάνουμε συνεδρίαση των συντονιστών και στις 2 θα πρέπει να ξεκινήσει η ακρόαση για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Έχουμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους Καταλαβαίνετε τις 3,5 ώρες συνεχόμενες. Ε, ζητώ την κατανόησή σας, θα δώσω το λόγο για ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, αλλά σας εκλεπαρώ ένα λεπτό καθένα, δύο λεπτά ο καθένας για να τα καταφέρουμε. Διότι η Επίτροπος Ρέντινγκ θα πρέπει να σας απαντήσει κιόλας. Δεύτερος γύρος λοιπόν ερωτήσεων σας παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε. Ο κύριος Άλβαρο. Uh, excuse me, Mrs. Gall. You... συγγνώμη, κυρία Γκάλ πρώτα. Συγγνώμη. Oh, Mrs. Gall. I, uh, I just want to, uh, to... Ήθελα απλώ να λάβω το λόγο, διότι αναφέρθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Επίτροπε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και είμαι βεβαία ότι θα κάνετε και κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει στον τομέα αυτό. Θα πρέπει άλλωστε. Είναι εκ των όνων ουκάνευ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω στη συζήτηση αφορά τις διάφορες φήμες που ακούγονται. Ε, Κυρία Γουίξτρομ, πρέπει να σας πω ότι αντίθετα με αυτά που μόλις μας είπατε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι άνοιξαν πάρα πολλά ε, καταφύγια προσφύγων, αστέγων, συγγνώμη, 600 νέα κέντρα αστέγων. Υπάρχει ένας ε, ειδικός ε, υπεύθυνο τη κυβέρνηση για, τις ε, περιοχές, ε, για τα καταφύγια αυτών αστέγων και κάποια κέντρα ψυχικής υγεία και όλα αυτά χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τους νέους νόμους τροποποιημένους και υπάρχει και νέα ποινικό, νόμο, νόμος, κυρία Γκάλ διακόπτει ο Πρόεδρος, και αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ε, επίθεση. Κυρία Γκάλα, αυτό είναι γύρω σε ερωτήσεων για την Επίτροπο. Καταλαβαίνω ε, ε, ότι έχετε κάτι να πείτε, αλλά απαντάτε στην Επίτροπο, ρωτάτε ερώτηση στην Επίτροπο. Απαντώ σε κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Ακούστηκε μια αδιανόητη κατηγορία εδώ. Γιατί λοιπόν άνθρωποι που αναφέρονται σε ζητήματα, και θα επανέλθω και στα της Επιτρόπου, δεν εξετάζουν τα γεγονότα και αρχίζουν να εξαπολύουν πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες χωρίς να εξετάζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πράγματι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαζόμαστε φορείς που πρέπει να εξετάζουν τι συνέβη, τα γεγονότα και να εξετάζουν και την νομοθεσία ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα και από αυτόν. Ευχαριστώ ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Άλβαρο, αλλά κυρία Γουίξερον, διαδικαστικό. Είναι πολύ σημαντικό διαδικαστικό ζήτημα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να ξεκινήσω συζήτηση με την κυρία Γκάλ. Ήμουν εδώ, όπω ήταν και η κυρία Γκάλ, για να συζητήσω με την Επίτροπο. Εκτιμώ το διάλογο με την Επίτροπο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι να μου επιτίθεται η Κίνγκα Γκάλ για το θέμα αυτό. Καλά κάνετε και ανοίγετε κέντρα αστέγων, αλλά δεν ε, δικαιολογεί ούτε διορθώνει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κονδύλια χαμένα για τους αστέγους. Εξαιρετικά είναι αυτά που κάνετε. Και δεν εκτιμώ το γεγονό να λαμβάνετε το λόγο και να δράτε ως μαριονέτα της κυβέρνησης Ορμπάν. Ο κύριος Άλβαρο, παρακαλώ. Καλώς βλέπουμε μια πρόγευση του τι μας περιμένει το απόγευμα. Έχει το ενδιαφέρον του και αυτό. Παρ' όλα αυτά, παίρνω το θάρρος επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής 8 έτη. Να πω ότι το θεωρώ πολύ κακό ως προσέλευση να έχουμε μόνο το 10% των μελών μας όταν έχει την Επίτροπος να μας μιλήσει για τόσο σημαντικά θέματα. Αυτό να το σκεφτεί κάθε ομάδα και η δική μου. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα δύο λεπτά που έχω, πολύ γρήγορα τρία θέματα. Εξτρεμισμός Ουγγαρία και προστασία δεδομένων. Για την προστασία των δεδομένων και τον κανονισμό κατανοώ την πρόθεση και γνωρίζω και την προεργασία. Εδώ και δύο χρόνια μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εκπρόσωποι συμφερόντων μου μιλούν για την ανανέωση της οδηγίας στην αναδιατύπωση. Ε, του κανονισμού μάλλον. Ε, είναι ενδιαφέρον, αλλά κοιτάξτε τι πρέπει να προσέξουμε. Τελικά, να μην βγει κάτι που να είναι ε, όχι καλές πράξεις, αλλά καλές προθέσεις. Ε, πολλά είναι τα ενδιαφέροντα, αλλά παραμένουν πάρα πολλά να διευκρινιστούν. Πολλοί ορισμοί νομικοί είναι πολύ δύσκολοι. 80% του κανονισμού τελικά μπορεί να αλλάξει μέσω εξουσιοδότηση ε, πράξεων, privacy by design, privacy by default, όντως του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Επίσης, είναι θεμητό να προστατεύουμε ε, τους πολίτες, αλλά δεν μπορεί εκείνοι που ε, χειρίζονται αυτά τα δεδομένα και ο επόπτης προστασίας δεδομένων ε, δουν μπροστά τους να ορθώνονται μεγάλα εμπόδια. Ας πούμε, επιχειρήσεις που να έχουν περιορισμούς ε, σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων, πάνω κάτω από 250. Επίσης, ε, δεν έχω χρόνο να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε. θα παρακαλούσα να έχουμε περισσότερο χρόνο, θα επιθυμούσα, ειδικά όταν είναι τόσο λίγα τα παρόντα μέλη, αλλά θα το ξανασυζητήσουμε. Έχουμε τόσο καλή και τόσο επαγγελματική σχέση που τι επόμενε εβδομάδε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και πάρα πολύ σύντομα γιατί γνωρίζω ότι ο χρόνο μου είναι περιορισμένο και θέλω να και άλλοι συνάδελφοι. Για την Ουγγαρία θα τα συζητήσουμε το απόγευμα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι έχω κι εγώ επιφυλάξει με εσά, ε, όπως και εσείς, τις διατυπώνω απλώ εντονότερα και ζητώ να προχωρήσουμε ε, σε προσφυγή βάσει του άρθρου 7.1. Ούτε εξέταση, δηλαδή να μην ζητήσουμε να διερευνηθεί αν έχουν παραβιαστεί. Πού είναι ο κόσμος. Κύριε Πρόεδρε, εκτό από εσά δεν υπάρχει κανένας άλλος σοσιαλδημοκράτης. Πού είναι οι πολίτες στη Γερμανία και θα τραγουδήσουν ένα τραγουδάκι που είναι πολύ γνωστό στη Γερμανία. Σοσιαλιστές μας προδώσατε. Που ομοιοκαταληκτεί και όλα στα γερμανικά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στην Επιτροπή μας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσουμε τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς σε τέτοια θέματα και στις αρμοδιότητες των αντιπροέδρων να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο για μένα σημαντικό που ε, είναι ε, η ε, κίνδυνοι των εξτρεμιστών ε, στην Ευρώπη. Αυτό αφορά και τους αναρχικούς στην Ελλάδα που στέλνουν ε, εμπριστικές επιστολές και βόμβες στο Δήμαρχο και αλλού, κουκουλοφόρους ας πούμε και ακροδεξιούς σε άλλες χώρες. Δεν έχω χρόνο και δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Συχώς πρέπει να σταματήσω. Ευχαριστώ κύριε Άλβαρο. Δεκτό τα όσα λέτε, έχετε δίκιο εμείς ως μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών έχουμε καθήκον να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε 60 μέλη, είμαστε γύρω στο, στους 20, εδώ δεν αρκούν όμως και ελπίζω στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών να υπάρχει η κατάλληλη εκπροσώπηση των πολιτικών ομάδων και να γίνει και το ίδιο σήμερα το απόγευμα όταν θα συζητήσουμε την κατάσταση στην Ουγγαρία ε, που θα κάνουμε και αυτή τη σημαντική ακρόαση. Κυρία Φλότρο. Ευχαριστώ. Δύο θέματα να θέσω και ένα σχόλιο να κάνω. Το πρώτο αφορά τους Ρωμά. Σωστά είπατε και θυμήσατε ε, ότι αντιδράσατε πάρα πολύ στεναρά μετά από τα γεγονότα του θέρους του 2010 στη Γαλλία και στη συνέχεια η Γαλλία άλλαξε την ομοθεσία της για την οδηγία της ελεύθερης κυκλοφορίας και πάρα πολύ καλά δράσατε και μπράβο σας. Ωστόσο, Πρέπει να σας πω ότι το 2011 στη Γαλλία είχαμε ακόμα περισσότερες απελάσεις ε, Ρωμά, Βουλγάρων και Ρουμάνων και συνεχίζουν οι πρακτικές. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών ε, να δημοσιεύονται. Δεν έχουν έρθει όλα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει σχόλια για το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει ακόμα όλα τα εθνικά προγράμματα, ε, δεν έχουν φτάσει στα χέρια σας ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τι πιστεύω και τι λέω, ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε αυτή την προσπάθεια συμπερίληψης στο Ρωμά, θα πρέπει να δούμε τις χώρες που διατηρούν τα προσωρινά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δείξετε εξίσου στεναρή στάση, γιατί είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματική ενσωμάτωση αυτών των προσώπων στην κοινωνία. Αν μπορείτε με τους συναδέλφους σας επιτρόπους να εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση για να είστε εξίσου δυναμικοί και στεναροί, θα ήταν πολύ καλά. Δεύτερο θέμα. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο δεν παρατηρεί στα κράτη-μέλη πρόοδο ε, για το σύστημα τη CIA για τα βασανιστήρια, ε, τις ανακρίσεις υπόπτων για τρομοκρατία κτλ, τις παράνομες αυτές δράσεις επειδή δεν ε, κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο πρότεινε μια έκθεση ε, συνέχειας στην έκθεση ΦΑΒΑ. Εσείς δηλώσατε πρόθυμοι να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εργασίας σας για το 2012 τι πρωτοβουλίες θα πάρετε, τι μέτρα θα πάρετε, γιατί από την έκθεση ΦΑΒΑ και μετά χάρη στην αιμονή και στην επιμονή δημοσιογράφων, δικηγόρων, μαρτυρίες, θυμάτων και ΜΚΟ έχουμε νέες πληροφορίες που οπωσδήποτε χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, ημών προσωπικά. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Αλφάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω κάποιες πτυχές και ελπίζω να μην υπάρξουν δυσάρεστε επιθέσει, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε και ζωντανά στο διαδίκτυο και είναι δυσάρεστα αυτά τα οποία επισήμανε ο συνάδελφο Άλβαρο. Είναι πολύ σημαντική συνεδρίαση και είναι ελάχιστοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ και για το γεγονός ότι πρόσεξε ιδιαίτερη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, την ε, έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα, στην οποία ήμουν εισηγήτρια και ε, μπόρεσα να μιλήσω και με τη Γενική Διευθύντρια Κνούτσεν επί του ζητήματος την περασμένη εβδομάδα. Τρεις ερωτήσεις, κυρία Επίτροπε. Στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αυτή τη στιγμή συζητάμε την πρόταση 7 κρατών μελών για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνα. Πρόκειται για μια πρόταση πολύ ενδιαφέρουσα για να βελτιωθεί η δικαστική συνεργασία, αλλά κατ' εμέ θα έπρεπε να αξιολογήσουμε κάποιες πτυχές λίγο καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόθεση να παρουσιάσει την πρότασή τη ούτως ή άλλως ε, και να κάνει και τι αξιολογήσει αντικτύπου οι οποίε θα ήταν απαραίτητες για μια τέτοια πρόταση. Δεύτερον, τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την ε, δικαστική κατάρτιση ε, με ιδιαίτερη αναφορά στο εργανομένο έγκλημα, στην νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Ε, σήμερα το πρωί στη Λιέγη συνελήφθη ένας δολοφόνος ο οποίος συμμετείχε σε μια οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος. Στην Κόζα Νόστρα. Και τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 για την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Δεν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την Ουγγαρία, κύριε Επίτροπη. Επιτρέψτε μου να αναφέρω. Η ξενοφοβική ρατσιστική ε, ε, συμπεριφορά εισβάλλει σε όλη την Ευρώπη. Και ακόμα και εδώ υπάρχουν βουλευτέ οι οποίοι καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση για ε, ρατσιστική συμπεριφορά. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω αυτή την ε, κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Γιάννουκα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή σας δέσμευση για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας ενημερώσατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στους 40 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που είναι οι φτωχότεροι και για τους οποίους χάρη στη βοήθειά σας ε, μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τους Ρωμά, αλλά δεν αφορά μόνο τους Ρωμά, αφορά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ένδυας. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ υποχρεώσεις και μια πολύ σημαντική ερώτηση επειδή διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο για να διευκρινίσετε το θέμα της ελεύθερης μετακίνησης και αναφέρετε και το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας για αυτούς τους φτωχότερους ανθρώπους μέσω του προγράμματος δράσης, έχετε να διαδραματίσετε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να διευκρινίσετε πώς ε, βοηθά η σχετική οδηγία όλους τους ανθρώπους ε, αυτούς που βρίσκονται στην Ευρώπη, ώστε αυτά τα ακραία φαινόμενα τα οποία αναφέρουν όλοι ε, και χρησιμοποιούν και ε, χειραγωγούν και τους Ευρωπαίους πολίτες και δημιουργούν πάρα πολύ σημαντικές εθνωτικές εντάσεις με την παραπληροφόρηση που κάνουν, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν θα συμβούν. Διότι για να καταπολεμήσουμε τι εξτρεμιστικέ τάσει θα πρέπει να δοθούν θέσει εργασία και να του δοθεί και ο λόγο αυτών των ανθρώπων. Όχι να μιλούν ε, κάποιοι εξ ονόματο κάποιων ομάδων, να έρθουν οι Ρωμά, οι ίδιοι φτωχοί ευθύ εξ αρχή και ε, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πρόγραμμα και να εφαρμοστούν τα προγράμματα και να παρακολουθούνται καταλήλω και από εκεί και πέρα θα έχουμε την κατάλληλη εικόνα των πραγμάτων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωση έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να γίνεται αντικειμενική ενημέρωση και να φροντίζουν να μην μαθαίνουμε μόνο τι ιστορικέ απόψει ε, κάποιων ανθρώπων που έχουν συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα, διότι από κάθε πολιτική πλευρά κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι στου οποίου αναφερόμαστε θα μπορούν να μα μιλήσουν οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εσείς να δείτε πώς ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τον εκτρομισμό στην Ανατολική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Στην Ουγγαρία οι δηλώσεις και οι απειλές σταμάτησαν πριν από μήνες όταν ο κύριος Ορμπάν επειδή εισήγαγε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά αλλά... Ε, υπήρξε και ο σχετικό νόμο που βοηθάει ιδιαίτερα. Η κυρία Ινέντφελτ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, έμαθα ότι κατόπιν αιτήματος των φιλελευθέρων την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια θα συζητήσουμε ένα ζήτημα για το οποίο αλληλογραφούσαμε το γραφείο σας ε, σε καθημερινή βάση στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, απορρίφθηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για θέματα προστασίας δεδομένων. Η απάντησή σας μέχρι τούδε ήταν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά εμεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να συζητήσουμε πώς μπορεί να διαθεροποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διασφαλίσει ότι στην Ευρώπη θα εφαρμόζονται μόνο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όχι η νομοθεσία τρίτων χωρών. Δεύτερον, για τα ομοφιλόφιλα ε, ζευγάρια και του γάμου ομοφιλοφίλων. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σε οικογενειακό δίκαιο, το οποίο και ισχύει. Αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμετέχει στη ε, βοήθεια για τις οικογένειες. Έχετε κάποιες πρωτοβουλίες για τις οικογένειες και το οικογενειακό δίκαιο και θα ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε το θέμα από αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Σάμσφασκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κόμμα του ε, Βίλτερς στην Ολλανδία είναι ξενόφοβο ε, και άνοιξε τώρα μία πύλη στο διαδικτύο που ενθαρρύνει τους πολίτες να καταγγέλουν για φαινόμενα και προβλήματα που έχουν με πολίτες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα και γίνεται και λόγος για απέλαση εργατών ε, από την Ανατολική Ευρώπη που ζουν στην Ολλανδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει τίποτα γι' αυτό. Το γνωρίζετε ότι συμβαίνει στην Ολλανδία και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 200.000 είναι οι εργαζόμενοι ε, στις κάτω χώρες με 1% μόνο ανεργία. Αυτά τα ξενόφοβα φαινόμενα είναι του παρελθόντος. Και ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει να τους βάζουν και το αστέρι στους Πολωνούς ε, εργάτες, όπως ε, στο παρελθόν. Αλλάζουν τα στοιχεία, τα ε, δεχόμενα, τα τα δεδομένα είναι αυτά καταστάσεις τύπου Εμβέρ Χόζα. Στο Βέλιο και στη Γερμανία απειλούνται πολιτικά κόμματα. Η αιρετική σκέψη σε κάποιες χώρες, σε πολλές χώρες ποινικοποιείται. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, η παράλογη ε, νομοθεσία στη Γαλλία που ποινικοποιεί τη δήλωση ε, ότι η ε, δολοφονία, οι των Αρμενίων και η δολοφονία από τους Τούρκους δεν ήταν γενοκτονία. Μα αυτά είναι επιχειρήματα, δεν χρειάζονται ε, ποινική δίωξη, χρειάζονται να αντικρουστούν με άλλα επιχειρήματα. Στην Ουγγαρία είδαμε τι έγινε το 2006 διαδηλωτές που γιόρταζαν την επέτειο του 56 κατεστάλησαν και έγινε λόγος για εξτρεμιστές. Εξτρεμιστές είναι οι πολιτικοί που θέλουν να απαγορεύσουν άλλα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί από όλες τις χώρες που ε, προσπαθούν να καταστήλουν την ελεύθερη έκφραση. Αναφερθήκατε στον έλεγχο για το χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων και πώς αυτός εφαρμόζεται. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η πολωνική κυβέρνηση πίστευαν ότι έχουν εξαίρεση. Ο κύριος Νταφ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων το έψαξε πρόσφατα και κατέληξε ότι είναι κενό γράμμα με βάση τα όσα είπε ένας εισαγγελέα που το έχει διερευνήσει. Δηλαδή η πολωνική και η αγγλική κυβέρνηση ε, ψεύδονται στους πολίτες όταν διαβεβαιώνουν ότι έχουν εξαίρεση. Και είμαι μέσα στα δύο λεπτά μου, πρόλαβα και τα είπα όλα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντινγκ έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και ραντεβού που δεν μπορεί να αλλάξει να λάβει. Αναβάλει, συγγνώμη. Τη δίνουμε το λόγο για να απαντήσει γιατί πρέπει να φύγει. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κι εγώ, Πρόεδρε. Η Ουγγαρία είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί το απόγευμα και στη συζήτηση αυτή πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να διαμορφώσει άποψη εάν θέλει να κινητοποιήσει τη διαδικασία βάσει του άρθρου 7. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει και το Κοινοβούλιο το ίδιο το άρθρο 7. Ε, προστασία των δεδομένων. Σίγουρα τώρα αρχίζει η συζήτηση, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες και στην ουσία. Είναι πολλά αυτά που έχει κανείς να πει, να συζητήσει, να αναλύσει και χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει πολύ εμπεριστατωμένη η εργασία και να αρχίσει τώρα. Για την ελεύθερη κυκλοφορία μίλησα ήδη και το θέμα των Ρωμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε βάσει των εθνικών ε, προγραμμάτων και σχεδίων δράσης ε, σε βάθος. Έγινε μια ερώτηση που δεν απάντησα ακόμα. Η έκθεση ΦΑΒΑ και τα ζητήματα της CIA μαζί με τη συνάδελφό μου Σεσίλια Μάλστρομ Έχουμε ασκήσει πολιτική πίεση στα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν την κατάσταση. Πολλά κράτη-μέλη κρύβονται πίσω από το απόρριτο και κάποια έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών ε, και δεν ε, είναι πρόθυμα να μας δώσουν αυτή την ενημέρωση. Το ζήτημα της κατάρτισης των δικαστών και της εκπαίδευσης ενισχύει τα όσα έχω κάνει. 700.000 δικαστές θα πρέπει να εκπαιδευτούν το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Η Eurojust να ενισχυθεί για τη συνεργασία των δικαστικών αρχών. Πώς το λέμε αυτό το Eurojust? Les procureurs. Ε, ε, ε, των εισαγγελέων. Ψάχνω τη λέξη στα αγγλικά. Οι εισαγγελείς λοιπόν πρέπει να συνεργάζονται. Και για το ξέπλυμα χρήματος και τέτοια θέματα ε, θα δουν νέες νομοθετικές προτάσεις να κατατίθενται σχετικά με τον ορισμό και τις ελάχιστες ποινές και πρόστιμα. Το Patriot Act μπορεί να είναι στην ημέρηση διάταξη για να συζητηθεί. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα διεθνούς δικαίου Εμείς θεωρούμε ότι βεβαίως και στην Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και όταν εμείς ζητούμε πληροφορίες για κάποια έκδοση, θα πρέπει βεβαίως να ανταποκρίνονται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εργαζομένων, εις βάρος των εργαζομένων στην Ολλανδία, Υπάρχει μια κοινή δράση. Εγώ μαζί με τον Επίτροπο Άντορ ε, κάναμε ένα διάβημα προς την Ολλανδική κυβέρνηση. Ευχαριστώ που είσαστε τόσο σύντομοι και τόσο περιεκτικοί και ε, ευχαριστούμε που καθίσατε τόση ώρα μαζί μας μέχρι τελευταία στιγμή της προσωρινής. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς για το χρόνο που μας έδωσαν. Σας ευχαριστώ όλους σας. Λοιπόν, συντονιστές, μην φύγετε. Έχουμε συντονιστές τώρα. Χρόνο δεν έχουμε για χάσιμο. Ευχαριστώ. Thank you.